να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Η πρωινή συνεδρίαση ήταν αρκετά κοπιώδης. Κάποιοι από τους βουλευτές φαίνεται να εξαντλήθηκαν, αλλά σίγουρα είναι εδώ όσοι έχουν αναλάβει ευθύνη των θεμάτων που θα εξετάσουμε. Θα προεδρεύσω εγώ μέχρι να έρθει η Πρόεδρος Σαρτόρη επίσης. Πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη, που βάσει του προγράμματος θα το συζητήσουμε περίπου για μισή ώρα, έχει να κάνει με τους προσανατολισμούς για τα ευρωπαϊκά επικοινωνιών. Να περάσουμε απευθείας στο θέμα. Θα μα παρουσιάσει το θέμα ο εισηγητή, ο κύριος Τοζενόφσκι, για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Τηλεπικοινωνιών και κατάργηση τη αποφαση αριθμο αριθμός 1336-97 και μετά θα ακούσουμε τι παρεμβάσει των σχεδόν εισηγητών και των υπόλοιπων συναδέλφων που θέλουν να παρέμβουν. Ο κύριος Τοζενόφσκι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως είπατε εσείς πολύ ωραία, Είμαι συντάκτης νομοδότησης για τα διευρωπαϊκά δίκτυα τηλεπικοινωνιών. Γενικά, καλωσορίζω πολύ την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί είναι ένα μέσο εξασφάλισης ε, της ευρυζωνικής ε, και της ψηφιακής ε, λειτουργίας του διαδικτύου. Και αυτό μπορεί να είναι ε, επίσης ε, κίνητρο για επενδύσεις ε, δημόσιες αλλά και ιδιωτικές. Χωρίς αυτή τη στήριξη κάτι τέτοιο θα ήταν αδύνατο ή θα ερχόταν πάρα πολύ αργά οπότε θα έπλητε την ανταγωνιστικότητα γενικώ. Υποδομές λοιπόν που έχουν προβλήματα ελλείψεις και ε, θα πρέπει αυτά να ξεπεραστούν, να επιληθούν. Και καλό είναι που το αναλαμβάνει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην το αφήσει στα χέρια ιδιωτών. τα μέσα θα πρέπει κυρίως να επικεντρωθούν στις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές, στις νησιωτικές περιοχές και σε θύλακες ε, ε, που ε, δεν καλύπτονται από ιδιωτικούς φορείς γιατί δεν τους ενδιαφέρει η κάλυψη και οι επενδύσεις εκεί. Σε ό,τι αφορά τις αστικές περιοχές δεν νομίζω ότι αυτό το μέσο είναι σκόπιμο να χρησιμοποιηθεί εκεί. Γιατί οι περιφέρειες και οι ιδιώτες επενδυτές ενδιαφέρονται να επενδύουν στις πόλεις γιατί τους αποφέρει αυτό κέρδος. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας και να είμαστε σε ε, αρμονία με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τα διευρωπαϊκά δίκτυα, ή υποδομές των τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να χρηματοδοτούνται όπου αυτό είναι απαραίτητο και σε κάθε περίπτωση. Και όπως σας είπα, είναι μια πρόταση η οποία συνοδεύεται και από τα απαραίτητα εργαλεία και μέσα για να φτάσουμε στους στόχους μας. Η αγορά του διευρωπαϊκού δικτύου τηλεπικοινωνιών θα πρέπει να ξεπεράσει όλα τα εμπόδια και να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα και την ανταγωνιστικότητα. Για να αναπτυχθούν αυτά τα δίκτυα θα πρέπει αυτό να βασίζεται σε συγκεκριμένους προσανατολισμούς όπως είναι ένα σύστημα ρητρών. Ε, τα δίκτυα και υπηρεσίε ε, που εγγράφονται σε αυτό το πλαίσιο είναι συγκεκριμένα μέτρα που θα πρέπει να επηρεάζουν θετικά την αγορά και να ε, καλύψουν τις ελλείψεις και τα προβλήματα που σήμερα γνωρίζουμε. Υπάρχει ένα ψηφιακό χάσμα σήμερα μεταξύ των πολιτών, ιδιαίτερα εκείνοι οι πολίτες που ζουν στην Ήπεθρο έχουν ε, λιγότερη κάλυψη θα πρέπει να καλυφθεί λοιπόν και η πεθρός και απομακρυσμένε και νησιωτικέ περιοχές. Ε, όλα αυτά θα μα επιτρέψουν να φτάσουμε σε ένα βασικό στόχο, Ακριβώ δηλαδή ε, την εύστοχη χρήση των πόρων για να ακολουθήσει η ανάπτυξη. στι λιγότερο ανεπτυγμένε περιφέρειες, εκεί είναι πιο χρήσιμη και πιο σημαντική η στήριξη και θα πρέπει να υποστηρίζεται κυρίως από τα διαρθωτικά ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής, εν προκειμένου. Επιπλέον, θα πρέπει η ψηφιακή αζέντα να φτάσει σε όλους τους πολίτες παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά λοιπόν. Η ψηφιακή στρατηγική για την Ευρώπη είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει όλα τα νοικοκυριά να έχουν τη δυνατότητα ε, τουλάχιστον έχουν πρόσβαση ε, σε διαδίκτυο με ταχύτητα 30 MB το δευτερόλεπτο μέχρι και 100 MB το δευτερόλεπτο. Ε, η επένδυση λοιπόν στην ευρυζωνικότητα γνωρίζει και ένα άλλο χαρακτηριστικό που ονομάζεται τεχνολογική ουδετερότητα. Τι είναι αυτό. Στην περίπτωση που παρέχονται υπηρεσίες σε μια συγκρίσιμη κλίμακα, θα πρέπει να ε, βεβαιωνόμαστε ότι δεν θα δρούμε με υποκειμενικό τρόπο ή με ελάχιστα αντικειμενικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν ορίζει ακριβώς ποιο τύπο τεχνολογίας θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Ποιος τύπος μάλλον. Και επίσης γίνεται λόγος για δυνατότητα χρήσης ε, δορυφόρων. κινητικότητα ε, και να υπάρχει παντού όσο γίνεται πρόσβαση σε ε, ευρυζωνικό διαδίκτυο και για μετακινούμενους ε, πολίτες. Για τη στρατηγική μας λοιπόν μπορούμε να συμφωνήσουμε με τις ιδέες, αλλά θέλω να ρωτήσω, με βάση ποια κριτήρια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέλεξε τα έργα για τα οποία ομιλεί στο κείμενό της, το οποίο αναφέρεται. Θα ενδιαφέρει αυτό δεχομένω και του συναδέλφους. Και περιμένω να ακούσω τις απόψεις και των συναδέλφων μας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να δούμε πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα μέσα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε ας πούμε, κάποιες ε, ε περιόδους καταστάσεις κρίσιμες, πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν ποιούνται από πυροσβέστες ή από τέτοιες υπηρεσίες και ε, να συνδυάσουμε όσο γίνεται τις προσπαθίες μας για να έχουμε προστιθέμενη αξία. Και εκεί χρειάζονται δημόσιες υπηρεσίες, δεν μπορούμε να περιμένουμε ο ιδιωτικός τομέας να αντικαθιστά ή να υποκαθιστά αυτές τις δημόσιες επενδύσεις που είναι τόσο κρίσιμες και τόσο χρήσιμες. Συμπερασματικά, θα ήθελα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς προτίθεται να ε, προωθεί σε αυτές τις υποδομές για τις ψηφιακές υπηρεσίες δεν έχω αρκετές διευκρινήσεις θα παρακαλούσα να το συγκεκριμένοποιήσετε στα πλαίσια του παρόντος κανονισμού πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος ε, από χρόνο να ενισχυθούν οι εξουσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής γιατί ε, ενδεχομένω να δημιουργηθούν προβλήματα και υποχρέωση ελέγχου από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έχουμε τις εξουσιοδότηση πράξης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό έχει πολύ μεγάλες εξουσίες ήδη σε ό,τι αφορά ε, την επιλογή ε, έργων δημοσίου συμφέροντος και θα πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου αντίστοιχο. Ελπίζω να είναι ο κανονισμός αρκετά ευέλικτος, να λαμβάνει υπόψη του δηλαδή ε, τις αλλαγές. Ε, θα πρέπει να υπάρχει νομική ασφάλεια, ασφάλεια δικαίου δηλαδή και ασφάλεια οικονομική εκτός από νομική. Όλα αυτά μέσω πρόθεσμα θα τα δούμε ε, για το πώς θα γίνεται ο έλεγχος να εξηγείται πολύ καλά η διαδικασία. Χρόνο έχουμε για να συντάξουμε τη γνωμοδότησή μας. Δεν πιέζει ο χρόνος και χαίρομαι ε, για την πολύ στενή συνεργασία που προσβλέπω να έχω με τους συναδέλφους για να λάβω υπόψη όλα τα σχόλια ε, σε αυτό το τομέα που είναι τόσο κρίσιμος όσο και χρήσιμος θα περιμένω λοιπόν να ακούσω τις απόψεις των συναντέλφων για ε, να δούμε όχι μόνο πώς θα προετοιμάσουμε ένα κείμενο, αλλά να κάνουμε και δημόσια κρόαση, που νομίζω ότι είναι πραγματικά πολύ ευστοχή ιδέα. Ακούστηκε η ημερομηνία 25 Απριλίου, είναι η επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας τότε για να μπορέσουμε να πάμε στην Ολομέλεια τον Ιούνιο. Λοιπόν, ανυπομονώ να ακούσω τις ιδέες σας και ευχαριστώ από τώρα τους ε, συνεργάτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε για την εισήγησή σας. Να ακούσουμε τώρα τι θα πει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σα έχουν τεθεί ήδη πολλά ερωτήματα. Υπάρχουν στην αίθουσα κύριοι σκιώδης συγκεκριτές, κυρία Τρότμαν. Ευχαριστώ, ε, αγαπητή Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο Τουζενόφσκι, τον εισηγητή μας, για το επικοδομητικό του πνεύμα. Εκ των προτέρων συνεννοήθηκε με τους Ε, εκτιμώ πάρα πολύ ε, τη στάση του και τα σχόλιά του που πραγματικά θέτουν το βασικό πλαίσιο της συζήτησης. Ε, ε, θα ήθελα καταρχάς να πω ότι σοσιαλιστές και δημοκράτες είναι υπέρ ενός προϋπολογισμού που να έχει πρικοδότηση αντίστοιχη με τις φιλοδοξίες μας. Η ψηφιακή στρατηγική είναι εμβληματική πρωτοβουλία και σχέδιο. Θα πρέπει να είναι όσο γίνεται καλύτερα ε, ζυγισμένη σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αν γίνεται να περιλαμβάνει και τα ευρωομόλογα. Σήμερα έχουμε μια πρώτη μόνο ανταλλαγή απόψεων, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, απλώς να θυμίσω ότι γίνεται λόγος για κατασκευή υποδομών. Δεν θα πρέπει όμως να ξεχνούμε το βασικό μας στόχο που είναι η μείωση του ψηφιακού χάσματος, της διαφοράς δηλαδή των πολιτών μεταξύ τους. Θα ήθελα Λοιπόν, εδώ να πω μερικές ιδέες ε, για να το σκεφτούμε από κοινού. Θα πρέπει ε, το ποσό που έχουμε ε, στη διάθεσή μας να πιάσει τόπο. Είναι 9,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Χρειάζεται να γίνουν επιλογές. Πώς θα κατανεμηθεί αυτό με μια κλίδα ανάμεσα στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την ηλεκτρονική υγεία που είναι υπηρεσίες και στην υποδομή. Χρειάζεται μια απαραίτητη ε, πολιτική ισορροπία ανάμεσα στις δημόσιες υπηρεσίες για ορισμένε περιοχές. Παράδειγμα, ε, θα, μπορούμε να έχουμε δωρεές εκεί και ΣΔΙΤ, ε, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Θα πρέπει να φροντίσουμε η στρατηγική αυτή να συνδεθεί με τα ταμεία συνοχής, τα οποία γνωρίζουν βαθιά μεταρρύθμιση κατά τα άλλα και αν ακούω αυτά που κυκλοφορούν, ε, διαπιστώνω ότι θα κληθούμε να κάνουμε ένα άθροισμα ε, των όσων χρειάζεται να χρηματοδοτήσουν αυτά τα ταμεία, αλλά τελικά δεν θα βγαίνουν οι λογαριασμοί στο, στο τέλος. Ε, είναι κρίσιμο αυτό και ευαίσθητο, ιδιαίτερα σε περιφέρειες που έχουν μείνει πίσω και χρειάζονται ιδιαίτερη στήριξη. Υπάρχουν και τα άλλα δίκτυα που πρέπει να υπάρχει μια διαλειτουργικότητα, ε, δίκτυα ενέργειας, δίκτυα μεταφορών. Ε, μπορούμε να το εξετάσουμε, ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες συνέργειες και συνεργασίες, αρχής γενομένης από τις πολιτικούς μηχανικούς κάποια στιγμή σε διάφορα προγράμματα, κατασκευών, έργα που μπορούν να γίνουν ταυτόχρονα για τις υποδομές, ε, μιλώ εδώ, και για τις διασυνδέσεις. Όλες οι πρωτοβουλίες θα πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται και να είναι συνεκτικές μεταξύ τους και συναφείς ε, σε ό,τι αφορά τον κανονισμό και βεβαίως λαμβάνοντας υπόψη και σεβόμενοι το πλαίσιο για τις τηλεπικοινωνίες και δι' ηλεκτρονικές. Κυρία Πρόεδρε, έχω μια ερώτηση και θα παρακαλούσα να μου απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, και την προσθέτω στις ερωτήσεις του εισηγητού. Αρκετά κράτη-μέλη έχουν κάποιες αισθητικές είδη για τις οπτικές ίνες και οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν διαφορετικές ευαισθησίες για το θέμα αυτό. Τι θα γίνει, ε, πώς θα συντονιστούν όλα αυτά και πώς θα επιταχυνθεί η κατάσταση και πώς θα συντονιστεί. Επίσης, πώς θα συνδεθούν με τα επιχειρησιακά σχέδια ε, των φορέων. Μα λένε ότι ένα έργο θα κινητοποιούνται τα κονδύλια. Ναι, αλλά αυτό μήπως οδηγήσει σε κατάσταση lock-in ορισμένων περιφερειών που θα είναι ένας παράγων που θα ε, μπλοκάρει τον ανταγωνισμό. Αυτός ο μηχανισμός δεν έχει ως προορισμό ε, να ε, χρηματοδοτεί αηφόρα και βιώσιμα έργα μόνο με χρήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Σήμερα οι ιδιώτες επενδύουν ε, σε έργα που δεν είναι απλώς βιώσιμα, αλλά είναι υπερβιώσιμα, ακόμα και σε αστικές περιοχές. Γιατί κάποια έργα που είναι αμφιβόλου κερδοφορίας ε, δεν τους ενδιαφέρουν για τους ισολογισμούς και για τα μερίσματα των μετόχων τους που είναι όλο και πιο απαιτητικοί. Και ε, το θέμα λοιπόν της δανειοδότηση και της χρηματοδότησης είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει αυτός ο μηχανισμός να παίξει σημαντικό ρόλο χρηματοδοτώντας ε, ε, έτσι ώστε αυτό να χρησιμοποιηθεί ως μια μαγιά και να προσελκύσει και άλλα κονδύλια. Για μια στρατηγική επενδυτική ε, μακράς διάρκειας και μακροπρόθεσμη. Γιατί 9 δισεκατομμύρια μπορούν να πολλαπλασιαστούν και να φέρουν και άλλα, αλλά ποτέ ε, δεν αρκούν για να καλύψουν το σύνολο της επικράτειας. Τι φρονεί γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν έργα που δεν χρειάζονται ε, δημόσια ε, στήριξη για να είναι βιώσιμα, αλλά εάν δεν έρθει μια ελάχιστη δημόσια στήριξη δεν πρόκειται ποτέ να ορθοποδήσουν. Ένας φορέα ε, τη αγορά στη χώρα μου ανακοίνωσε στου μετόχους του ότι θα μειωθεί το μέρισμα γιατί θα χρησιμοποιηθούν αυτά τα χρήματα για επενδύσεις. Εγώ το θεωρώ θετικό αυτό, αλλά θα δούμε τι ανταπόκριση θα έχει. Ε, τώρα, για την ε, πολιτική προστασία και ασφάλεια που ανάφερε και ο εισηγητή, το Κοινοβούλιο πάντα ενδιαφέρεται γι' αυτό, ιδιαίτερα για το ραδιοφάσμα και σε μια ρύθμιση που πρόσφατα εγκρίθηκε υπάρχει ειδική διάταξη που λέει ότι θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη υπηρεσίε επίγουσα αντίδραση και πολιτική προστασία. Αυτά είναι τα λίγα σημεία που θα ήθελα να σα αναφέρω και το υποβάλλω στην κρίση σα, στη σοφία σα, αλλά και στι ικανότητε Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ εκ των προτέρων την Επιτροπή και τον εισηγητή για τι απαντήσει. E Ευχαριστώ. Είναι μακρύ ο κατάλογο των ερωτήσεων, ε, λέω προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, το λέω γιατί θα χρειαστούμε πολύ συγκεκριμένε απαντήσει. Ο κύριος Σόκμαν. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τον εισηγητή, τον κύριο Τασνόφσκι, για την εξαιρετική παρουσίασή του, η οποία αποτελεί μια πολύ καλή βάση για όλους μας που συμμετέχουμε σε αυτή την εργασία. Είναι βασικό να κοιτάξουμε το περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε. Ήδη έχουμε αναπτύξει μία νέα πολιτική ε, φάσματος και ιδίως όσον αφορά τη, τα ε, στοιχεία που διακινούνται μέσω κινητών τηλεφώνων και ζητάμε πολύ περισσότερα από αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ένα άλλο θέμα στα πλαίσια αυτά είναι ότι αυτός είναι ένας τομέας ε, ο οποίος προχωρά πάρα πολύ γρήγορα στις κοινωνίες μας και ε, χρειάζονται ε, χρηματοδοτήσεις οι οποίες δεν είναι εύκολος και γι' αυτό ε, λόγω κόστους δεν μπορούν να γίνουν και μεγάλες ε, νέες εγκαταστάσεις και μόνο στην κοινική τηλεφωνία για να έχουμε την ε, ε, ταχύτητα των 30 MB και 100 MB πολύ πριν το 2020 θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι δεν πρέπει να καταρτήσουμε στόχους οι οποίοι μακροπρόθεσμα θα μας, θα μας εμποδίσουν διότι μιλάμε για το 2020 λες και είναι αύριο αλλά έχουμε 8 χρόνια μπροστά μας οπότε εάν κοιτάξουμε που ήμασταν πριν 8 χρόνια το 2004 δηλαδή Δηλαδή, όπου η τεχνολογία ακόμη ήταν πολύ διαφορετική και δεν είχαμε δει να εμφανίζονται τόσα θέματα που θεωρούμε δεδομένα σήμερα σχετικά με τις υπηρεσίες μεταδόσεως στοιχείων όπου ε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ο τεράστιος όγκος διακινήσεως στοιχείων των οποίων θεωρούμε δεδομένο φοβάμαι όπως σας είπα ότι αν μιλάμε για το 2020 θέτουμε στόχους, το πράγμα που είναι καλό ε, για του χρόνου, αν μιλάμε για το 2013. Αλλά από τώρα μέχρι το 2013 και από εκεί ως το 2020 θα συμβούν πάρα πολλά και είμαι βέβαιος ότι οι στόχοι τους που οποίους κατήρτισε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ξεπεραστούν από την πραγματικότητα. Δηλαδή η πραγματικότητα προχωρά πολύ πιο γρήγορα σε αυτό το τομέα από την νομοθεσία. Θέλω λοιπόν να παρακαλέσω τον εισηγητή να το σκεφτεί και να ε, κοιτάξει οι στόχοι που έχουν τεθεί ε, και ο τρόπος με τον οποίο θα τους επιτύχει να είναι βιώσιμοι. Ε, και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροφή να μας εξηγήσει ποιοι είναι οι στόχοι για το 2020, δηλαδή εάν πιστεύουν ότι υπάρχουν εφικτές αυτές ε, προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν οι ε, στόχοι αυτοί το 2020 αν μιλάμε για ένα συγκεκριμένο αριθμό μεταδόσεως μεγαμπάιτ παραδείγματος χάρη πρέπει ναι μεν να είμαστε θαραλέοι αλλά πρέπει να είμαστε και φιλόδοξοι διότι διαφορετικά θα προγραμματίζουμε και θα προγραμματίζουμε να μείνουμε στην τέταρτη ή στην πέμπτη θέση. Ενώ θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα είμαστε πρωταγωνιστές σε αυτό το τομέα. Ένα άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε ε, τα κριτήρια για να μπορέσουμε να καλύψουμε ε, τις προποθέσεις του Ταμείου Συνοχής και άλλων ταμείων ας μιλάμε για επενδύσεις οι οποίες ε, θα είναι ε, περισσότερες ε, από εάν δεν είχαμε αυτούς τους πόρους γιατί οι εμπορικές επενδύσεις είναι ταχείες και χρησιμοποιούνται σε όλη την Ευρώπη αλλά όχι σε όλες τις περιοχές όλης της Ευρώπης. Οπότε θέλουμε να στηρίξουμε την εξέλιξη της, του μεγαλύτερου όγκου στοιχείων πολύ περισσότερο από ό,τι θα μας εξασφάλιζαν εμπορικές επενδύσεις. Και γι' αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε οι επενδύσεις τις οποίες θα διευκολύνουμε με αυτόν τον τρόπο να, να γινόντουσαν ούτως ή άλλες. Δηλαδή είτε επενδύαμε εμείς είτε όχι. Διότι ξέρουμε ότι στις μεγάλες μας πόλεις ε, υπάρχει το ευρυζωνικό σύστημα με μεγάλη ταχύτητα και ε, εδώ κανονικά συζητάμε ε, για τα προβλήματα που προκύπτουν όταν προτρέχουν οι εξελίξεις στις μεγάλες πόλεις. Επίσης ε, η διαχωριστική γραμμή στο ψηφιακό σύστημα γιατί προχωρούν πολύ πιο γρήγορα οι εξελίξεις στις πρωτεύουσες των χωρών μας αλλά μετά ε, λαχανιάζουν οι άλλες περιφέρειες να ε, προλάβουν και υπάρχουν και άλλα θέματα που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Αυτό λοιπόν με οδηγεί σε ένα τρίτο θέμα και ένα συμπέρασμα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Διότι δεν πιστεύω ότι εκτός εξαιρετικών περιστάσεων όπου τίποτα δεν θα συνέβαινε όπου δηλαδή ε, πρέπει να είμαστε πολύ φιλόδοξοι στις, ε, στα μεγάλα αστικά κέντρα, στις πρωτεύουσες ότι πρέπει κανείς να απευθύνεται ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, θα πρέπει να απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κάθε φτωχιά περιοχή, περιοχή με λιγότερη χρηματοδότηση, η οποία δεν έχει την οικονομική εξέλιξη την οποία θα επιθυμούσαμε και κατά κανόνα αλλά επίσης και με όλες τις ε, εξαιρέσεις που μπορούν να προκύψουν ε, θα πρέπει να φροντίσουμε τα χρήματα αυτά να μην αποδοθούν στις μεγάλες αστικές περιοχές όπου ούτως ή άλλως θα υπάρξουν επενδύσεις. Παρακαλώ λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μου πει επί του θέματος αυτού πώς αυτό μπορεί να τυπωθεί. Διότι εάν χρησιμοποιούμε τους πόρους αυτούς για τα πάντα δεν θα μπορέσουμε να είμαστε τόσο φιλόδοξοι όσο θα θέλαμε εάν ξοδέψουμε όλα τα χρήματα και δεν μας μείνει τίποτα. Ευχαριστώ. Με συγχωρείτε, αλλά ο χρόνος τρέχει και περνά πολύ γρήγορα. Δεν μου ζήτησε ε, να επέμβει κανείς άλλος σιώδης εισηγητής. Ο κύριος Κρόιτσμαν, η κυρία Χάιντς Ντότερ θέλουν να επέμβουν σας παρακαλώ να είσαστε πάρα πολύ σύντομος γιατί ο προλαλής σας δεν σεβάστηκε το χρόνο του. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, χθες ε, η εφημερίδα Handelsblatt μιλά για ε, γρήγορα δίκτυα που δημιουργούν νέες ελπίδες και δημιουργούν γρήγορες δυνατότητες μεταδόσεως για να αυξηθεί η σημασία τους. Δηλαδή όπου υπάρχει το σωστό επενδυτικό σχήμα υπάρχουν Μεγάλε μεγάλες επενδύσεις και δεν χρειάζεται κανείς να βοηθηθεί από ευρωπαϊκούς πόρους διότι καλύπτεται από τους ιδιώτες επενδυτές. Αλλά αυτό που μας απασχολεί είναι περιοχές οι οποίες δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσες για τις τηλεπικοινωνίες ή υπεθρος παραδείγματος χάρη, όπου και εμείς θα πρέπει να στρέψουμε το βλέμμα μας και υπάρχει μία προστιθέμενη αξία μέσω του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών και με το μέσο Connecting Europe προσπαθούμε να δώσουμε μία νέα όθηση. Αλλά αυτό δεν έχει άμεση σχέση με το Connecting Europe αλλά ουσιαστικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για το τηλεπικοινωνιακό σύστημα της Ευρώπης όπου προσπαθεί κανείς να προωθήσει την ανάπτυξη της Ευρώπης οικονομικά. Θα πρέπει λοιπόν να κοιτάξουμε τις άλλες περιοχές της Ευρώπης οι οποίες ε, έχουν προχωρήσει πάρα πολύ ε, διότι ε, οι μεν προχωρούν γρήγορα και άλλες υστερούν πάρα πολύ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να δώσει τη δυνατότητα να έχει κανείς πρόσβαση σε ορισμένα μέσα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτό είναι σημαντικό στο διάλογο μεταξύ κρατών μελών. Επίσης οι χρήστες πρέπει να έχουν εμπιστοσύνη στο ασφαλές διαδίκτυο και θα πρέπει να πατάξουμε τις παράνομες δραστηριότητες. Όσον αφορά τους στόχους όπου επενδύονται ε, ε, στα ενεργειακά δίκτυα θα πρέπει να ξεχωρίσουμε ότι το διαδίκτυο είναι πιο σημαντικό για τους χρήστες και θα πρέπει να προωθηθεί. Ε, επίσης πρέπει να αναφερθούμε στο πιο βασικό θέμα που είναι τα ευρυζωνικά δίκτυα διότι χωρίς αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί καμία από τις υπηρεσίες που θέλουμε. Πρέπει να προχωρήσουμε πολύ και να υπάρξουν οι αναγκαίες δομές ακόμη και αν πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν και δεν υπάρχει τίποτα. Γνωρίζω το πρόβλημα από την ε, περιοχή μου Rheinland Pfalz όπου αυτή τη στιγμή δεν έχουμε ευρυζωνικά δίκτυα και εδώ το μέσο Connecting Europe μπορεί να μας βοηθήσει. Είναι βασικό όμως παρόλες τις καλές ε, προθέσεις να διερευνήσουμε εάν επιτυγχάνουν οι επενδύσεις, εάν υπάρχει μία μετακίνηση των πληθυσμών ή αν χρειάζεται κάτι άλλο τέτοιο στο μέλλον και, να, και επιπλέον αν υπάρχουν εναλλακτικέ τεχνολογίες. Δεν χρειάζεται πάντοτε να πρόκειται να ε, είναι σταθερά να, ε, ε, χρειάζεται πάντα να είναι σταθερά δίκτυα, αλλά θα πρέπει να βρεθούν και πιο ενδιαφέρουσε λύσεις για ορισμένες περιοχές, διότι εδώ μιλάμε μόνο για την επίτευξη ε, των, των ζωνών των 30 και 100 MB, πράγμα το οποίο μπορεί να αλλάξει στο μέλλον και είναι κρίμα να περιοριστούμε η εις ε, τις οπτικές Πρέπει να ε, αναρωτηθούμε εάν σε ένα χωριό στην ε, στην Ήπεθρο δεν θα βοηθηθεί κανείς καλύτερα με ε, μία δομή με λιγότερα μεγαμπίτ η οποία θα κοστίζει και λιγότερο και θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της ε, συγκεκριμένης περιοχής. Προσβλέπω στη συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η, κυρία Χάιντς Ντότερ θέλει να επέμβει. Eh, eh, Ευχαριστώ τους συναδέλφους για τις ε, τοποθετήσεις ε, και τα όσα μας είπαν. Έχω μια ερώτηση. Ευχαριστώ ε, πολύ ε, για τις προτάσεις της στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί πραγματικά την απασχολούν και αυτά τα θέματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ε, στην Ήπεθρο. Εγώ όμως δεν έχω πιστεί τελείως από τις μεγάλες επενδύσεις στα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, εάν και κατά πόσο αυτό είναι πανάκια ή εξυπηρετεί κάθε σκοπό. Εμείς έχουμε εμπειρίες από δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ήπεθρο σε κάποιες περιφέρειες της Ένωσης που δεν είναι πάντα θετικές. Χρειάζεται εκτός από την κινητή τηλεφωνία ένα χερσαίο δίκτυο και μάλιστα υπόγειο δίκτυο με οπτικές ίνες, ιδιαίτερα εκεί ε, που οι περιοχές είναι ιδιαίτερα ρεοκατοικημένες. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ, ε, κυρία Πρόεδρε. Πολύ ενδιαφέρον το έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και πολύ ε, χρήσιμο ε, για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορούμε να λύσουμε πολλά προβλήματα έτσι. Ανησυχούν πολλοί συνάδελφοι όμως, όχι μόνο εγώ και η κυρία Μανδουρέλ και άλλοι, για τις ε, τεχνολογίες που θα μας επιτρέψουν στο μέλλον να φτάσουμε στους στόχους μας. Εμείς που μπήκαμε στην Ένωση το 2004, ε, καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες για ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και ε, υπογράψαμε και συμβάσεις περίοδου 4 μέχρι 7 ετών. Έτσι έχει πραγματικότητα, αλλά αλλάζει σήμερα και έχουν ξεπεραστεί αυτές οι συμβάσεις. Ε, και θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παίζει σήμερα περισσότερο και μεγαλύτερο ρόλο στη χάραξη των μεγάλων κατευθυντήριων γραμμών σε αυτό το τομέα. Να υπάρχει δε και δυνατότητα συμμετοχή σε συζητήσει για τις νέες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να βελτιωθεί η μεταφορά δεδομένων σε όλες τις περιφέρειες και η προσέγγιση και η πρόσβαση στις πληροφορίες. Ευχαριστώ. Ε, για να απαντήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ελπίζω να είναι σαφής και περιεκτική μέσα σε τρία λεπτά η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Uh, um, Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω για τα καλά σας λόγια, για την υποδοχή ε, που επιφυλάξατε στην πρόταση είναι ε, πραγματικά στην καρδιά της ε, πρότασης του 2020 του Πρόεδρου Παρόσου αλλά και του Επιτρόπου Ευχαριστώ τον συγητή, τους σκιώδης εισηγητές και όλους τους υπόλοιπους βουλευτές. Είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω σε οποιασδήποτε άλλες ερωτήσεις, αλλά προς το παρόν να περιοριστώ σε αυτές που κάνατε σήμερα. Συμφωνούμε απολύτως ότι η πρόταση ως έχει σήμερα φιλοδοξεί να μειωθεί το ψηφιακό χάσμα αλλά και το κόστος της ψηφιακής τεχνολογίας. Αυτή είναι η ψηφιακή ατζέντα η λεγόμενη και ο στόχος της. Γι' αυτό σχεδιάζουμε όλα αυτά να τα ε, υλοποιήσουμε μόνο, όχι μόνο από το μέσο ε, Connecting Europe, αλλά ένα σύνολο, ένα χαρτοφυλάκιο και με άλλα μέτρα πολιτικά και δημοσιονομικά, τα οποία ε, αυτό τον καιρό υλοποιούνται και θα συνεχίσουν να υλοποιούνται και στο μέλλον. Ε, μπορεί να υπάρξει συμπροματικότητα με τα διορθωτικά ταμεία στο βαθμό που ο κανονισμός του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου δεν τα περιορίζει. Αναθεωρήσαμε την πρόταση ακριβώς για αυτό τον σκοπό και το λόγο. Εξαρτάται βέβαια αυτό σε μεγάλο βαθμό από την προεθυμία των μεμονωμένων κρατών μελών αλλά και του Κοινοβουλίου να Ε, δει τι γίνεται με την ευρυζωνικότητα και πώς αυτή λειτουργεί ε, μέσα στα διαφορετικά ταμεία. Η σημερινή πρόταση ως έχει επιτρέπει κάποιες συνεργασίες και δεν επιτρέπει κάποιες άλλες. Εμείς φροντίσαμε, προτείνουμε να βελτιστοποιήσουμε την κατάσταση ακριβώς επειδή είναι περιορισμένη οικονομική πόρη ε, που μπορεί να διαθέσει ο δημόσιος τομέας της επενδύσης εκεί. γνωρίζουμε απολύτως και έχουμε πλήρη επίγνωση του γεγονότος ότι δεν είναι εύκολο να καθορίσει κανείς ακριβώς τη συμπεριφορά και τη στάση ιδιωτών επενδυτών εταιριών τηλεπικοινωνιών όταν παίρνουν αποφάσεις για τις επενδύσεις τους. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ευρυζωνικότητα, η δική μας παρέμβαση επικεντρώνεται στην υποστήριξη των ε, πρωτοβουλειών ε, καθώς αυτές αναπτύσσονται και είναι διαθέσιμες. Δηλαδή, η πρόταση δημιουργεί ένα χώρο για να λάβουν τα κράτη-μέλη την ε, ηγετική αυτή προσπάθεια, όπως κάνει αυτό τον καιρό η Γαλλία, για να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες σε περιφερειακό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων, κοινοτήτων, σε άλλα κράτη-μέλη. Είναι πολύ ουσιαστικό κάθε φορά που επιτρέπει ένα έργο τη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, εμείς τη διευκολύνουμε. Έτσι λοιπόν στην πρόταση για το μέσο και τη διευκόλυνση Connecting Europe θα δείτε και αναφερομένη την πρόταση ε, και τη δέσμευση ότι εμείς κυρίως επικεντρωνόμαστε στα χρηματοδοτικά μέσα. Η επιλογή λοιπόν των έργων θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών και από τις ΣΔΙΤ, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, γιατί είναι πρόθυμοι να προτείνουν και να προωθήσουν. Εμείς ε, ζητήσαμε να υπάρχει κάποια ευελιξία και να βοηθούμε ε, τις δημόσιες αρχές ε, να εγκαθιστούν δίκτυα ευρυζωνικά κυρίως στην Ήπεθρο και επίσης θέλουμε να ε, δοθεί συνέχεια σε κάποιες καλές πρακτικές που ήδη ε, υφίστανται ε, σε κάποια μέρη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα μπορούσαν να αντιγραφούν και να μεταφερθούν αλλού. Ξέρουμε ότι αυτός ο τομέας κινείται με ταχύτητα τους ρυθμούς και αναπτύσσεται. Γι' αυτό οι κατευθυντήριες γραμμές στο διευκόλυνση Connecting Europe προτείνουν κάποια ευελιξία. Ξέρουμε ότι υπάρχει ανάγκη για έλεγχο και ε, για συμμετοχή και των πολιτικών στη λήψη των αποφάσεων, αλλά μια πρόταση με πάρα πολλές λεπτομέρειες ε, θα ε, ήταν πάρα πολύ άκαμπτη, τελικά θα κατέληγε μη λειτουργική και μη εφαρμόσιμη και απολύθωμα σε τελική ανάλυση υπάρχει ένα επίπεδο φιλοδοξιών και ένα επίπεδο αξιοπιστίας. Από το, ακούμε από την αγορά, ε, οι στόχοι που πρότεινε η Επίτροπος κυρία Κρούς, ε, νομίζω βρίσκουν ανταπόκριση και η αγορά είναι πρόθυμη να τη σκεφτεί. Έτσι όπως ε, έχει η πρόταση, και από το δημοσιονομικό κανονισμό είναι η εξής. Για να χρησιμοποιηθούν δημόσια κονδύλια θα πρέπει να υπάρχει αδυναμία του ιδιωτικού τομέα. Δηλαδή στόχος δεν είναι να παραγωνιστεί ο ιδιωτικός τομέας και ε, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων έτσι και έχει ένα κανόνα που λέει ότι δεν μπορεί να υποκαταστήσει ε, τις ιδιωτικές επενδύσεις. Σε ό,τι φορά τις υπηρεσίες, αν θέλετε να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφό μου για να σας απαντήσει εκείνος. Με συγχωρείτε για ένα λεπτό αν γίνεται, γιατί πραγματικά έχει περιοριστεί ιδιαίτερο ο χρόνο μα, Πρέπει και εμεί να ακολουθήσουμε το ρυθμό των εργασιών μα. Όχι παραπάνω από λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα απαντήσω πολύ συγκεκριμένα στην ερώτηση που μου κάνατε. Για τις υπηρεσίες έχουμε τρία διαφορετικά κριτήρια για ε, τη ψηφιακή έλλειψη. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει αρκετή οριμότητα στις περιφέρειες για τις υπηρεσίες αυτές. Σήμερα είναι σε πιλωτικό στάδιο. Θα πρέπει να οριμάσουν αρκετά για να επιλεγούν και επίσης να είναι σε ένα, στο επίπεδο της ανάπτυξης, της υλοποίησης ήδη. Αυτοί είναι οι τρεις λόγοι που μας οδήγησαν να επιλέξουμε τα διάφορα έργα που ε, βλέπετε στο παράρτημα της πρότασής μας. Ε, πρέπει να σας πω επίσης ότι ο κατάλογος αυτός δεν είναι ε, οριστικός, είναι ανοιχτός, μπορούν να προσθεθούν και άλλα. Θα μπορούσαμε σε συνεργασία με τους νομοθέτες να προσθέσουμε και άλλα έργα ή να αφαιρέσουμε στον βαθμό που αυτό χρειάζεται. Και τελειώνω λέγοντας το εξή στη μητρική μου γλώσσα, που είναι τα σουηδικά. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ήπεθρο που ρώτησε η κυρία Άντερς Ντότερ. Είμαι βέβαιος ότι θα τις βοηθήσει αυτή η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα έλεγα να καθιερώσουν μια καλή πρακτική. Οι εκπρόσωποι της Επιτροπής γραπτώς να απαντούν ε, πολύ συγκεκριμένα στις ερωτήσεις που έχουν γίνει. Δηλαδή, Εάν δεν θέλετε ότι δεν προλάβατε να το γράψετε, να μας γράψετε τις απαντήσεις σας, τόσο το καλύτερο. Να δώσω τώρα το λόγο στον ε, κύριο το Ζενόφσκι, εφόσον θέλει οπωσδήποτε να απαντήσει, αλλιώ καλύτερα να αποφύγουμε και την δεύτερη παρέμβαση από εκείνον. Ωραία λοιπόν, μπορούμε να κλείσουμε με, αυτά, με αυτές τις παρατηρήσεις. Είπες ότι δεν θες το λόγο. Ε, Κοιτάξτε, δύο αντιδράσεις. Συμφωνώ απολύτως με την κυρία Τροτμάν. Είναι πολύ σημαντικό να εκτιμήσουμε το οικονομικό εύρος της πρότασης αυτής για να μπορούμε να δούμε και τι βάρη θα επιφέρει. Και θα συμφωνήσω απολύτως και με τον κύριο Πάκερ, είμαι ειδικό πληροφορικής, αντεπάγγελμα. και όταν ήμουν φοιτητής Ήταν υπέροχε οι σπουδέ που έκανα τότε εμένα, αλλά έχουν ξεπεραστεί προπολού. Οι εξελίξει είναι ραγδαίε. Σε λίγα μόλι χρόνια έχουμε πάει πολύ μακριά. Σα ευχαριστώ λοιπόν και αναμένω διακαώ την συνεργασία με του συναδέλφου. Σα ευχαριστούμε. Γνωρίζετε το χρονοδιάγραμμα των προθυσμιών. Όλα τα υπόλοιπα γραπτό. Επόμενο σημείο στην εμμυρίσια διάταξη. Τρίτο πρόγραμμα για την ε, υγεία η συγκήτρια Μπαντία Κουτσέ, ε, η κυρία Μπαντία Κουτσέ, την οποία είναι πολύ σύντομη γιατί είμαστε ε, ήδη αργά. Ναι, Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομη, θα σα ακούσω. Αλλά νόμιζα ότι πρώτα ήταν η άλλη έκθεση για την επιγραμμική διανομή οπτικοακουστικών έργων. Πρόεδρε, με ακούτε. Στη δική μου ημερησία διαταξή λέει πρώτα την επιγραμμική διανομή και όχι την υγεία. Α, ναι, ναι, δικιά σας είναι και η προηγούμενη. Ναι, ναι, έχω δύο εκθέσεις. Όχι, την υγεία να πείτε πρώτα. Ωραία. Γνωρίζετε ότι είναι γνωμοδότηση ε, για, για παντάει για το άλλο θέμα η κυρία ε, Μπαντία Κουτσέτ. Ε, η επιγραμμική διανομή οπτικοακουστικών έργων είναι της Επιτροπής Πολιτισμού. Την είχε ο κύριος Ένσιου ε, αρχικά. Μετά ανέλαβα εγώ την έκθεση αυτή και θα ήθελα να σας πω ότι αυτό που έκανα ήταν να συνεχίσω τη δουλειά του κυρίου Ένσιου και να προσθέσω και κάποιες δικές μου ιδέες. Οι βασικές ιδέες της έκθεσης είναι ο κατακαιρματισμός της επιγραμμικής διανομής και της αγοράς. Υπάρχουν τεχνολογικά εμπόδια, περίπλοκες διαδικασίες αδειοδότησης και χρειάζεται συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να φτάσουμε προς μία ενιαία ψηφιακή αγορά. Επίσης θα πρέπει να δίνεται περισσότερη προσοχή στη βελτίωση ε, των πλατφορμών επιγραμμικής διανομής για να γίνονται σεβαστά τα πνευματικά δικαιώματα και τα οπτικοακουστικά ε, στην επιγραμμική διανομή πλατφόρμες διανομής, δηλαδή τεχνολογικές εταιρείες, πάροχοι υπηρεσιών ε, και ε, οργανώσεις κοινωνίας των πολιτών. Επίσης, υπάρχει ανάγκη να ε, αμείβονται σωστά οι Ε, παραγωγή ή δημιουργή και θα πρέπει να γίνουν μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βρεθούν απαραίτητοι μηχανισμοί για να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι το Γραφείο Εναρμόνισης Εσωτερικής Αγοράς που πρόσφατα ανέλαβε προστασία των ε, δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας προσφέρεται να κάνει αυτές τις μελέτες και έτσι θα αποφύγουμε ε, περιττή επικάλυψη οργανισμών και θα μπορέσουμε να χειριστούμε καλύτερα τους οικονομικούς πόρους. Και τέλος, τονίζεται η σημασία του προγράμματος Δημιουργική Ευρώπη για να διανέμεται επιγραμμικά το προϊόν της οπτικοακουστικής ε, βιομηχανίας. Έτσι συνεισφέρουμε και στην ε, κοινωνική συνοχή. Αυτές είναι οι βασικές ιδέες της γνωμοδότησης και με χαρά θα ακούσω τις προτάσεις και τις απόψεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Μαντία Κουτσέ. Μας είπε ήδη πολλά, σε πολύ λίγο χρόνο, αλλά μας έδωσε πολλά στοιχεία. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Κυρία Άντιστότερ. Ευχαριστώ. την εισηγητρία η κυρία Μπαντία Κουτσέ για την παρουσίασή της. Προφανώς ε, θεωρούμε ότι όσο περισσότερο περιεχόμενο υπάρχει στο διαδίκτυο, τόσο πιο πολύπλοκο γίνεται το πώς θα δενέμεται μέσα από το διαδίκτυο. Θα προσκαλέσει, ελπίζουμε, η έκθεση αυτή του ιδιωτικού φορείς να συνεργαστούν διότι αυτή η μέθοδος εργασίας μπορεί να επηρεάσει την ουδετερότητα του δικτύου ή την διανομή πληροφοριών στο δίκτυο. Μπορεί να υπάρξουν δηλαδή επιπτώσεις, σοβαρές επιπτώσεις για την εδαφικότητα, την περαιτέρω ανάπτυξη της ενιαίας αγοράς και της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Ήθελα λοιπόν να μάθω τι σκέφτεται η εισηγήτρια σε σχέση με το θέμα αυτό. Άλλες ε, παρεμβάσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Ανδρό, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην πράσινη βιβλό, που δίνει συνέχεια στη στρατηγική για την πνευματική διοκτησία, όπως ξεκίνησε τον Μάιο του 2011, περιλάβαμε όλες τις ενισφορές, ήδη και στο διαδίκτυο, διατίθενται προς τους πάντες και όλο το κοινό. Έχουμε πάνω από 220 αιτήματα και απαντήσεις. Με πολλούς ε, από τους κατόχους δικαιωμάτων να συμμετέχουν και ετοιμάζεται νομίζω έκθεση για την επόμενη χρονιά με δημόσια ακρόαση προς το τέλος του καλοκαιριού. Το αργότερο τον Οκτώβριο. Με συγχωρείτε, αλλά ως προς την ερώτηση που τέθηκε... Από την, κατά την προηγούμενη παρέμβαση, νομίζω ήταν μια ερώτηση για την ε, εισηγήτρια, έτσι. Ήταν, ε, ζητήθηκε η άποψη του εισηγητή, της εισηγήτριας ή ήταν σε σχέση με την πράσινη βιβλό. Δεν είμαι βεβαίω. Όχι, αφορά την πρόταση της εισηγήτριας. Για την εισηγήτρια ήταν η ερώτηση. Ολοκληρώσατε. Πολύ ωραία. Κυρία Μπαντία Κουτσέ, Έχετε λίγα λεπτά. Ευχαριστώ για τα σχόλιά σας. Για την ερώτηση που ε, κατάλαβα ότι ήταν προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να σας δώσω και εγώ τη γνώμη μου. Έχει αποδειχτεί πλέον ότι είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε μια απάντηση. Πώς διατηρούμε αυτή την ισορροπία από τη μια τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, αλλά και από την άλλη την πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, την επικοινωνία και τον πολιτισμό που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Δεν ξέρω πόσα χρόνια συζητούμε όλα αυτά τα θέματα σε πολλές επιτροπές και είναι σημαντικό να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και τώρα θα πρέπει να γίνει αυτή η ακρόαση πολύ γρήγορα και χαίρομαι που την αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γιατί θα πρέπει να βρούμε μια λύση όλοι οι ενεχόμενοι σε συνεννόηση. Οι καταναλωτές, οι παραγωγοί, οι δημιουργοί, οι πάντες, όσοι ενέχονται σε αυτή την προσπάθεια, καλούνται να συνεργαστούν για να βρούμε μια λύση. Εκείνοι που δημιουργούν, ε, λοιπόν, ε, έχουν κάποια δικαιώματα, αλλά και το κοινό, το ευρύ κοινό θέλει πρόσβαση. Ε, αυτή τη μάχη πρέπει να δώσουμε όλοι από κοινού. Ευχαριστώ πολύ. Θεωρούμε ότι ολοκληρώνει τη συζήτηση. Η προθεσμία είναι στις 7 Μαρτίου δεν την υποβολή τροπολογιών και η ψηφοφορία θα γίνει στις 24 Απριλίου. Και τώρα ο λόγος και πάλι στην κυρία Μπαντία Ικουτσέ για το πρόγραμμα για την υγεία, το τρίτο πρόγραμμα πολιτικού δράσης για την υγεία, είναι το επόμενο θέμα που θα μας παρουσιάσει. Έχετε πέντε λεπτά αυτή τη φορά για την παρέμβασή σας. Σας ε, ζητώ συγγνώμη που σας πίεσα τόσο πολύ προηγουμένως. Δεν θα τα χρειαστώ καν. Θα είμαι και πάλι πολύ σύντομη αυτό το πρόγραμμα ε, της υγείας στην υπηρεσία της ανάπτυξης έρχεται μια στιγμή που είναι μεγάλες οι προκλήσεις που συνδέονται με την παγκοσμιοποίηση, την κρίση στην οικονομία αλλά και τη γύρανση των κοινωνιών μας. Το πλαίσιο της στρατηγικής για το 2020 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λανσάρει αυτό το θέμα υγεία στην υπηρεσία της ανάπτυξης για περισσότερη έρευνα, για διατήρηση των συστημάτων υγείας, για βελτίωση της υγείας των πολιτών και να προστατευτούν από τα δυσυνοριακά προβλήματα και απειλές για την υγεία τους. Ωστόσο, είναι πολλές οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνδέονται και με άλλους τομείς που έχουν σχέση με την ε, υγεία και δεν τα αξιοποιεί αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχει ανάγκη να αξιοποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα για να γίνεται έρευνα στην υγεία συντονισμένη ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι καταγερματισμένη. Έτσι θα είναι πιο βιώσιμη και πιο ανεπτυγμένη η ίδια η έρευνα. Επίσης, θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανισότητες και μεταξύ τομέων του πληθυσμού και μεταξύ περιφερειών για την υγεία. Τα μεταναστευτικά ρεύματα έχουν φέρει ασθένειες που ήταν μέχρι τώρα απλώς στις αναπτυσσόμενες χώρες και τώρα υπάρχουν και είναι καθημερινή πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή δράση εκεί, όχι μόνο θα αντιμετωπίσουμε τις ανάγκες της Ένωσης, αλλά θα βελτιώσουμε και το βιωτικό επίπεδο στις αναπτυσσόμενες χώρες και έτσι ε, θα βοηθήσουμε και τις οικονομίες τους. Επίσης, χρειάζεται να συνεργαζόμαστε στην υγεία για την ανάπτυξη με μια εμβληματική πρωτοβουλία, νέες ε, δεξιότητες για νέες θέσεις εργασίας, new skills for new jobs. Ιδιαίτερα ε, αυτά που ονομάζουμε θέσεις εργασίας της λευκής μπλούζας, δηλαδή ε, οι εργαζόμενοι στην υγεία και στις κοινωνικές υπηρεσίες. Το υγειονομικό προσωπικό που ε, απασχολεί σήμερα 20 εκατομμύρια περίπου πολιτών και έχει ε, μεγάλες ε, δυνατότητες ανάπτυξης γιατί αντιστρέφεται η πληθυσμιακή πυραμίδα, γυρνάει ο πληθυσμός μας δηλαδή το πρόγραμμα αυτό μπορεί να μην είναι ερευνητικό πρόγραμμα, αλλά θα πρέπει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που δίνουν η καινοτομία και οι νέες τεχνολογίες για να ε, αναπτυχθεί η αποτελεσματικότητα και η αποδοτικότητα. Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε τις προόδους που έχουν γίνει ε, στις τεχνολογίες που βασίζονται ε, στο ραδιοφάσμα και ε, το ε, ίντερνετ ε, των στόχων που είχε παρουσιάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πέρυσι. Θα ήθελα και πάλι να ακούσω τις απόψεις σας για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο, λόγ, ο λόγος στην πρώτη σχέδιση, γιατί την κυρία Τζόρνταν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια για την εισήγηση την οποία έκανε. Όντως το έγγραφο αυτό είναι απαραίτητο λόγω της κρίσεως και λόγω της γυράνσεως της κοινωνίας αλλά θέλω να προσθέσω ότι ασχολούμαστε επίσης και με την ε, τις κλιματικές αλλαγές και πρέπει να δούμε τι επιπτώσεις έχει και ο τομέας αυτός. Είναι πολύ σωστό ότι το θέμα αυτό ε, δεν πρέπει απλούστατα να εξεταστεί από τη σκοπιά της ε, υγείας των ανθρώπων αλλά ε, από την σκοπιά επίσης και της γενικότερης εξέλιξης. Και εδώ μιλάμε για την περίοδο μέχρι το 2020 και θα υπάρχει λίγο λιγότερο υγειονομικό προσωπικό, πράγμα το οποίο θα, θα προκαλέσει μία πρόκληση σχετικά με την γύρανση του ευρωπαϊκού πληθυσμού και πρέπει να δούμε πώς θα εμποδίσουμε οι άνθρωποι να αρρωσταίνουν συχνά. Ένας άλλος τομέας που θα μας απασχολήσει είναι ε, επίσης ε, ε, και οι διευκολύνσεις που θα πρέπει να υπάρχουν και οπότε θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε δημιουργήσουμε ε, μία προστιθέμενη αξία ε, και ε, την συνέργεια και για να υπάρχει ένα συνδυασμός με άλλους τομείς όπως τα διαρθρωτικά ταμεία ή ο ορίζον 2020 οι προτάσεις ε, για ε, τροποποιήσεις και οι τροπολογίες που έχουν υποβληθεί δεν με βρίσκουν πάντοτε σύμφωνοι ε, ιδίως όσον αφορά τους πιο ευπαθείς πληθυσμούς και την αλληλεπίδραση με τους, τις κινήσεις των κρατών μελών. Θα πρέπει εδώ να εξετάσουμε τους τέσσερις στόχους στόχους οι οποίοι καταρτίζονται στο πρόγραμμα αποτελούν ε, προτεραιότητες και πρέπει να είναι ισοσχελισμένοι. Πολύ σωστά το είπε η ε, η συγγήτρια διότι είπε ότι δεν χρειαζόμαστε μόνο ένα πρόγραμμα για την έρευνα και έρευνα και ενοτομία, αλλά πρέπει όλα να συνάδουν και να εξελιχθούν από κοινού και να μπορέσουν να προβλεφθούν διάφορες ενέργειες οι οποίες προβλέπονται στο νομοθετικό κείμενο όπου ζητάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χρηματοδοτήσει άμεσα χωρίς να προβλέπεται καν στο ετήσιο πρόγραμμα ε, ε, επενδύσεων αλλά επειδή τα ποσά είναι σημαντικά είναι κάτι που θα πρέπει να ξανασκεφτούμε πριν δεχθούμε ότι θα χρηματοδοτούνται προγράμματα χωρίς δημόσιο διαγωνισμό και ε, αν ε, ναι θα πρέπει τουλάχιστον να υπάρχουν κριτήρια τα οποία θα πρέπει να καθοριστούν δηλαδή το έγγραφο αυτό πρέπει να είναι σαφέστερο και θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις απόψεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πράγμα το οποίο δεν έγινε στην αρχή και γι' αυτό εγώ θα επιθυμούσα η ανεξαρτησία των μη κυβερνητικών οργανώσεων να είναι πιο σαφής και να είναι σαφές ότι πρέπει να είναι πολιτικά ανεξάρτητες. Σας ευχαριστώ. Αν δεν υπάρχουν άλλες επενδύσεις, το λόγο έχει ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, ο κύριος Ζεώ. Το όνομά μου είναι Ρόμπερτ Σόλτεκ και εγώ θα παρέμβω εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ πολύ για την δυνατότητα που δόθηκε στην Επιτροπή Ήτρε να εκφράσει τη γνώμη της επί της προτάσεως. Είμαστε σε επαφή με την εισηγήτρια και μπορέσαμε ήδη να συζητήσουμε ορισμένες προτάσεις. Ελπίζουμε δε ότι θα διευκρινιστούν και διάφορα θέματα. Όσον αφορά το σχέδιο γνωμοδότησης που έχει καταρτιστεί, Συμφωνούμε ότι το πρόγραμμα αυτό πρέπει να εξεταστεί από την οπτική γωνία της γενικότερης στρατηγικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη του 2020 και ο τίτλος το διεκηρύσει αυτό, δηλαδή πρέπει να δούμε πώς θα συμβάλλουμε ή στην ανάπτυξη και επίσης ε, στο γεγονός ότι ε, πρέπει να υπάρχει υγεία για να μπορέσει να υπάρξει ανάπτυξη. Τονίζουμε ότι Όσον αφορά τις ε, ε, ασθένειες που έχουν σχέση με τη φτώχεια και την εγκατάλειψη ε, γεωγραφικά μπορεί να υπάρχει μία εφαρμογή σημαντική του προγράμματος αυτού διότι είναι περιοχές οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο γενικότερο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως θα μπορέσουν να υπάρξουν δηλαδή αλληλεπιδράσεις και ευχαρίστως θα δεχθούμε τις τροπολογίες που αναφέρονται σε τις ε, ε, θέσεις εργασίας σε γραφεία που συνάδουν ε, με την, τις δικές μας στην Επιτροπή όσον αφορά το πρόγραμμα υγείας και τον ορίζοντα για την έρευνα του 2020 υπάρχει ε, μία κατανομή εργασίας. Είμαστε μικρότερο πρόγραμμα από αυτό της έρευνας και ο στόχος μας και η φιλοδοξία μας δεν είναι να γίνει έρευνα για την έρευνα μόνο αλλά να προωθηθεί η έρευνα στα κράτη-μέλη μέσω του υπάρχοντος συστήματος και ε, της συνεργασίας με τα κράτη-μέλη. Όσον αφορά τις παρατηρήσεις της κυρίας Τζόρνταν Τσίζελ την διαβεβαιώνω ότι δεν ε, υπάρχει καμία πρόταση η οποία θα γίνει ή θα υιοθετηθεί χωρίς να εφαρμοστούν οι κοινοτικοί κανόνες για δημοσιονομικά θέματα κατά τρόπον ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μία χρηστή διαχείριση των πόρων των φορολογουμένων και όλα αυτά θα διαχειρίζονται από μία επιτροπή. Δηλαδή οι δράσεις με τα κράτη-μέλη θα γίνονται κατόπιν προκηρύξεως ενός ε, διαγωνισμού. Δεν είναι δηλαδή απλώς προτάσεις για εφαρμογή προγραμμάτων, απλώς θέλω να σας εξηγήσω πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Αλλά αν θέλετε μπορούμε να μιλήσουμε και διμερώς και θα βρούμε την άκρη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η συγγήτριά μας θέλει να απαντήσει. Παρακαλώ. Ναι. Θέλω μόνο να ευχαριστήσω για τη συνεργασία την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την κυρία Τζόρνταν για τα καλά της λόγια. Και βέβαια θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα αυτό και να εργαζόμαστε έτσι ώστε η έκθεση να συνεισφέρει έτσι με ενδιαφέροντα τρόπο ε, στο πρόγραμμα υγεία στην υπηρεσία της ανάπτυξης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Τροπολογίες θα πρέπει να μας έρθουν έως τις 7 Μαρτίου το μεσημέρι. Ο κύριος Κέλλη. Με συγχωρείτε. Ήθελα να ζητήσω το λόγο προηγουμένως για την επιγραμμική διανομή οπτικοστικών έργων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Μπέλετ, ο σχεδόν εισηγητής, είναι στη Βερμανία για συγκεκριμένη επίσκεψη σήμερα. Οπότε θα ήθελα να διαβάσω κάτι εκ μέρους του. Διότι χάθηκα λίγο με τις αλλαγές στη σειρά της ημερησία διάταξης. Μπορώ. Κυρία Μπαντία Ικουτσέ. Εγώ, evidentemente, no εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα προφανώς να διαβάσει ο κύριος Κέλλη τη σελίδα που του έδωσε ο κύριος Ιβο Μπελέτ. Αλλά μπορούμε να το δούμε και διμερώς. Δεν χρειάζεται τώρα να επιβαρύνουμε τη διαδικασία. Αν θέλετε, εμένα δεν με πειράζει. Αλλά είναι θέμα που τελείωσε και έχουμε πάει σε άλλο και τώρα έχει να διαβάσει ένα κείμενο άλλου συναδέλφου. Σας προτείνω να το δούμε διμερώς και να τελειώνει η υπόθεση. Εντάξει, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, διότι θεωρητικά έχει λήξει η συζήτηση με την ε, Επιτροπή, με τις παρεμβάσεις όλων. Μπορούμε να συμπεριλάβουμε στα πρακτικά τον, ε, την παρέμβαση του κυρίου Μπέλετ και μετά τα συζητάτε μεταξύ σα. Είναι απλούστερο. Νομίζω θα ήταν καλοδεχούμενη αυτή η λύση αν και εσεί μπορείτε να συμφωνήσετε. Αφήστε μα λοιπόν τη γραπτή συνεισφορά τη γραμματεία του κυρίου Μπελέτ και θα τα δει η συγγήτρια και τα, συζητάτε μετά, τα συζητάνε μεταξύ τους. Περνάμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Σημείο 18. Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση τη παραποίηση απομίμηση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωση και των κρατών μελών της αφενός και αφετέρου της Αυστραλίας, του Καναδά, της Ιαπωνίας, της Δημοκρατίας του Κορέας, του Μεξικού, του Μαρόκου, της Νέα, Ζηλανδίας, της Σιγκαπούρη, της Ελβετίας και των Πολιτειών. Ο λόγο στην κυρία Άντερ Δότερ, Αμέλη Άντερ Δότερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους και όλους τους που με βοήθησαν ειλικρινά και ουσιαστικά μέχρι τώρα. Αυτή η εμπορική συμφωνία γνωρίζετε ότι στοχεύει στη κατάργηση, καταπολέμηση της παραπίσης και απομίμησης και ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει διαπραγματευτεί αυτό το θέμα το 2007 μέχρι το 2010. Έχουν γίνει ήδη εμπορικέ ε, διαπραγματεύσεις, αλλά εν πλήρη αδιαφανία. Επανειλημμένα καταφέραμε να περάσουμε ψηφίσματα για να βελτιώσουμε την πρόσβαση στα έγγραφα και τη διαφάνεια τους ε, δύο τελευταίους μήνες. σε πολλά κράτη-μέλη δόθηκε μεγάλη προσοχή σε αυτή τη συμφωνία ε, με πολλές διαμαρτυρίες, με πολλές αντιστάσεις και πολλές συζητήσεις. Και εμείς στο Κοινοβούλιο έχουμε κινήσει την προσοχή ε, πολλών. Έχουμε λάβει και εσείς θα έχετε λάβει πολλές ε, επιστολές, τηλεφωνήματα, email από πολίτες της Ένωσης που ανησυχούν για τις επιπτώσεις αυτής της συμφωνίας. Εμείς ως ε, θεσμικό όργανο και ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή θα έπρεπε τουλάχιστον να δούμε ε, τι γίνεται στη βιομηχανία και τι επιπτώσεις έχει στη βιομηχανία η δική μας ε, παρέμβαση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε την περασμένη εβδομάδα να εκδώσει δελτίο τύπου που αφορά τα μελήματα και τις ανησυχίες των πολιτών και τώρα έχουν προσφύγει και στο δικαστήριο το οποίο θα αποφανθεί ε, εάν όλα αυτά είναι σύνομα. Μπράβο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επέλεξε αυτή τη δικαστική οδό, αλλά ε, τίθενται και πολλά ερωτήματα ε, ως προς τη βιομηχανία που δεν μπορούν να απαντηθούν ε, με τέτοια απόφαση δικαστική. Παράδειγμα, οργανισμοί τηλεπικοινωνιών επανειλημμένα ανησυχούν και αγωνιούν και λέγουν ότι στη συμφωνία τα κράτη ε, υποχρεούνται ρητά να συνεργάζονται με ιδιωτικές εταιρείες. Και αυτό ε, έχει θορυβήσει ε, τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών ότι θα διασαλευτεί η ουδετερότητα και η ανεξαρτησία των επιχειρήσεων. Η πλατφόρμα δηλαδή για τους χρήστες και για τις εταιρείες θα πρέπει να είναι ανοιχτή και ουδέτερη. Επίσης, ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, ανησυχούν στην Ευρώπη ότι θα έχει αρνητικές επιπτώσεις και για τις μελλοντικές τους δραστηριότητες αυτό το σύστημα. Πολλές έννοιες στη συμφωνία αυτή. Επίσης, χρειάζονται προσοχή, διότι δεν είναι παραδοσιακές στην ευρωπαϊκή νομολογία. Δηλαδή, δεν είναι φαινόμενα που γνωρίζουμε ήδη από το παρελθόν. Έχουμε ερωτηματικά. Για την ερμηνεία ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι θα σημαίνει αυτό για τη βιομηχανία. Ο κόσμος ανισχύει, φοβάται, προβληματίζεται. Τι θα γίνει με τις τρίτες χώρες. Μπορεί να εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία σε άλλες χώρες και αυτό θα οδηγήσει σε εμπόδια εμπορικά. γιατί μπορούν να μπουν διάφορα φίλτρα και διάφορα εμπόδια ε, στο διαδίκτυο και αυτό να εμποδίζει ευρωπαϊκές εταιρείες να δραστηριοποιούνται σε ε, αλλοδαπές αγορές. Όλα αυτά τα ερωτήματα δεν έχουν απαντηθεί συγκεκριμένα, δεν έχουν ελεγχθεί. Παράδειγμα, πώς επηρεάζει τις τηλεπικοινωνίες αυτή η συμφωνία ή τι επιπτώσεις μπορεί να έχει στην ε, καινοτομία και στις προσπάθειες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Έχει προκύψει τώρα μια νέα κατάσταση ιδιαίτερη λόγω της προσφυγής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο δικαστήριο και η δική μας δουλειά του Κοινοβουλίου ως θεσμικό οργάνου αλλάζει και έχει κάπως παραγωνιστεί. Ε, μας έχουν λίγο εκτοπίσει. Και δεν θα έχουμε μάλλον την ευκαιρία να αποφανθούμε ως θεσμικό όργανο, ως κοινοβούλιο, μετά την απόφαση του ε, ΔΕΚ. Και το μέλλον αβέβαιο θα εξαρτηθεί πολύ από αυτά που θα αποφασίσει αύριο η Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου, ΙΝΤΑ. Εγώ πιστεύω θα ήταν κρίμα εάν σταματούσε εδώ η πολιτική συζήτηση που έχει ακριβώς γεννήσει τόσο ενδιαφέρον στα κράτη-μέλη από πλευρά των πολιτών και χρειάζεται να συζητηθεί εφόσον ανησυχούν τόσο πολλοί οι πολίτες. Ενδεχόμενη λύση θα μπορούσε να είναι η δική μας Επιτροπή να ζητήσει μελέτη που δεν έχει ακόμα ανατεθεί για το πώς θα μπορούσε να επηρεάσει αυτή η συμφωνία την ενδοτερότητα του δικτύου ή την εξέλιξη και ανάπτυξη των επιγραμμικών υπηρεσιών. Αυτό θα μπορούσαμε να το κάνουμε μέχρι να βγάλει το δικαστήριο την απόφασή του να αναθέσουμε μια τέτοια μελέτη. Και κάτι άλλο που είναι σημαντικό και για μένα και για τους σκιώδης ε, γιατί παρακολουθούμε και τις εργασίες ε, στην Επιτροπή Εξωτερικού Εμπορίου, ε, ΙΝΤΑ, Διεθνού καλύτερα. Ακούσαμε ότι εκεί θα κάνουν μάλλον μια προσωρινή έκθεση για να διατηρηθεί η δημοκρατική συζήτηση, να μην κλείσει είναι και αυτό ένα θέμα που μπορούμε να εξετάσουμε και να βοηθήσουμε κι εμείς ε, προς την κατεύθυνση αυτή. Από τη σκοπιά της βιομηχανίας. Θα μπορούσε ενδεχομένω και η νομική επιτροπή Γιούρι να αναμειχθεί και να πει ότι το Κοινοβούλιο επιθυμεί να παρακολουθήσει την εξέλιξη στο Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για να μην ε, βγούμε εκτός ε, αυτής της διαδικασίας. Πολλά μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο, αλλά δεν έχουμε ακόμα βεβαιότητα για το πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Θα σας τηρούμε όλους ενήμερους για το πώς εξελίσσεται η υπόθεση και ε, περιμένω με χαρά να ακούσω τα σχόλια των συναδέλφων. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα, πολύ μεγάλο και θα μας απασχολήσει ακόμα σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την εισηγησή σας. Ο κύριος Ντεάντζελης, σκιώδης εισηγητής. Παρακαλώ. Άντζελης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχω εκτιμήσει ιδιαίτερο το έργο τη εισηγήτρια. Θαυμάσια έκθεση. Και άριστη βάση για τη συζήτησή μας. Δεν θα μακρηγορήσω για το πόσο ενδιαφέρον είναι το θέμα αυτό για το κοινό. Ξέρετε τις όλες τις συζητήσεις για την Συμφωνία Άκτα και ξέρετε το φάσμα που καλύπτουν όλες αυτές οι... όλα αυτά τα ζητήματα. Τώρα, ένα καθοριστικό ζήτημα. Το κατά πόσον θέλουμε να κάνουμε την Ευρώπη κοινωνία της ε, πληροφορίας και ενημέρωσης. Το να έχουμε κανόνες για το περιεχόμενο ε, στο διαδίκτυο θα πει ότι θα περάσουμε στις ψηφιακές επικοινωνίες και την ε, οικονομία της γνώσης και θα πρέπει να επηρεάσουμε τη λειτουργία τους. Ε, σε πολλά κράτη-μέλη υπήρξαν κινητοποιήσεις, διότι υπάρχουν κανόνες ε, για την διακυβέρνηση του διαδικτύου στη Συμφωνία Άκτα. Επηρεάζει λοιπόν τον κυβερνοχώρο, όπου οι πολίτες συνήθως έχουν ελεύθερες σχέσεις μεταξύ τους, χωρίς περιορισμούς. Όμως η Συμφωνία Άκτα είναι πάνω απ' όλα μια συμφωνία κατά τις παραποίηση και απομίμησης. Ε, δεν ε, θέλει να επιτρέπει την ε, διανομή των παραποιημένων προϊόντων που μπορεί να επηρεάζουν την επιβίωση ολόκληρων αγορών εργασία. Και βεβαίω είναι και επικίνδυνα για του καταναλωτέ. Για το θέμα λοιπόν αυτό, το να γίνει κάτι που εδώ και πολύ καιρό το αναβάλαμε, δηλαδή να χτυπήσουμε τι διεθνεί μαφίε που χειρίζονται την διακίνηση παραποιημένων εμπορευμάτων. Μην ξεχνάμε ότι και σε προηγούμενε θητείε το Κοινοβούλιο αυτό είχε εγκρίνει εκθέσει πρωτοβουλία και νομοθετικέ προτάσει που ήθελαν να ορίσουν αυστηρότερου κανόνε για την κατάσχεση εμπορευμάτων. Νομοθετικέ ε, διατάξει και ε, νέε νομοθετήματα και διάφορε μορφέ συνεργασία. Στο Συμβούλιο, βέβαια, οι διαπραγματεύσει ξεπεράστηκαν από τι ίδιε τι εξελίξει. Αναφέρομαι στην οδηγία ΕΠΕΝΤ 2, που θα μπορούσε να μα δώσει πολλέ ιδέε για το πώ να διορθώσουμε κάποια από τα σημεία τη Συμφωνία Άκτα που μπορεί να μα ικανοποιούν. Πάντω, ο αγώνα κατά τη παραποίηση και τη απομίμηση είναι κάτι σημαντικό και θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποια συγκεκριμένα ωφέλη θα μπορούσαμε να αποκομίσουμε μια συμφωνία που δεν λαμβάνει υπόψη τι ε, χώρες όπως η Κίνα ή η Ινδία. Και πώς ο ΟΗΕ, ο ΠΟΕ ή άλλοι διεθνείς οργανισμοί θα καλύπτουν την ισχύ της συμφωνίας αυτή. Ε, πιστεύω ότι ο αγώνας κατά των ε, παραποιημένων ή ε, εμπορευμάτων είναι κάτι που να το δούμε με έναν τρόπο βελτιωμένο. Δηλαδή θα πρέπει εδώ να κυρώσουμε μια επιλογή μας. Θα πρέπει να γεφυρώσουμε τις διαφωνίες και τις αντιφάσεις για να έχουμε μια θέση πιο ενιαία. Η συμφωνία αυτή είτε θα απορριφθεί είτε θα εγκριθεί, γιατί αν δούμε το άρθρο 27 της συμφωνίας, η επιγραμμική πειρατεία δείχνει ότι υπάρχουν, για την επιγραμμική πειρατεία δείχνει ότι υπάρχουν ζητήματα και μεθοδολογικά και ουσίας. Τα πνευματικά δικαιώματα μπορεί να θεωρηθούν και στα πλαίσια του εμπορικού δικαίου ως ποινικά κολάσιμα κάποιες φορές ε, με κάποιες ενέργειες. Και έτσι επηρεάζεται και το ηλεκτρονικό εμπόριο. Εδώ λοιπόν είναι μια... έχω να κάνω μια συζήτηση που δεν αποτελεί νέο στοιχείο για την Ευρώπη και θίγει διαφορετικές ευαισθησίες και συμφέροντα. Η συμφωνία λοιπόν άκτα δεν επιλύει απολύτως το πρόβλημα της παραποίησης, αλλά παρεμβαίνει και σε μια συζήτηση που έχει να κάνει με την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο. Σε μία συμφωνία τέτοιου εύρους, το Ευρωκοινοβούλιο δεν μπορεί να παραμείνει απλώς θεατής. Πρέπει να δούμε τι διαβουλεύσεις, τι συζητήσεις θα διοργανωθούν με το κοινό, με την κοινωνία των πολιτών, τι μελέτες αντικτύπου υπήρξαν σήμερα για να έχουμε μια ενιαία θεώρηση του θέματος αυτού. Αλλά φαίνεται ότι όσα έγιναν ως τώρα ήταν απλώς μια υφολογική άσκηση. Και μάλιστα σε μια περίοδο που η ευρωπαϊκή εξοπιστία έχει πληγεί ιδιαίτερως. Επί της ουσίας νομίζω ότι η συμφωνία δείχνει ότι οι υπηρεσίε στο διαδίκτυο θα πρέπει να διακυβερνώνται από συγκεκριμένου κανόνε. Όμω, οι πάροχοι των υπηρεσιών δεν μπορούν να παρακολουθούνται απλώ δικαστικά. Η ισχύουσα νομοθεσία δεν έχει προβλέψει βέβαια κάτι σχετικά. Ούτε τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται παρκώς με την νέα συμφωνία για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων στο διαδίκτυο θα πρέπει να έχουμε μια πιο προσεκτική εξέταση ώστε να βασιστούμε σε συγκεκριμένε γνώσει και στοιχεία. Ούτε ο ιδιωτικό βίο δεν προστατεύεται με του κανόνε που, που προτείνονται. Όμω και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα αποφανθεί για την συμβατότητα τη συμφωνία με τα θεμελιώδη δικαιώματα όπω ε, τα θεσπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάντω, ο αρμόδιο επίτροπο, βάσει των τελευταίων ειδήσεων που έχουμε, επανέλαβε ότι η ΑΚΤΑ είναι μια συμφωνία που θέλει να ανυψώσει τα διεθνή πρότυπα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Δικαιώματα που θα έπρεπε να καλύπτονται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μετατροπή του πώς αντιλαμβανόμαστε τους παρόχους υπηρεσιών στο διαδικτύο. Όμως εδώ δεν φαίνεται να έχει ληφθεί επαρκώς υπόψη η Ευρωπαϊκή Νομοθετική σκοπιά. Η συμφωνία αυτή θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει και την πολιτική μας τοποθέτηση στο θέμα αυτό. Για την παραποίηση των εμπορευμάτων Βεβαίω και δεν θα πρέπει να επιτραπεί στους μεγάλους παραγωγούς παγκοσμίω να διαχέουν και να διακινούν παραποιημένα εμπορεύματα. Όμως αυτό που αναζητούμε εδώ και χρόνια είναι μια ενιαία θεώρηση για την ε, πειρατεία στο διαδίκτυο. Τι εμπορικές επιπτώσεις μπορεί να υπάρχουν και τι κοινωνικές φθορέ μπορεί να προκληθούν. Με βάση τη απόφαση λοιπόν το δικαστήριο, το Ευρωκοινοβούλιο θα πρέπει να, ε, ε, να ενισχύσει το κύρος του τοποθετούμενο και σε σχέση με αυτή τη συμφωνία που τελικά δεν προστατεύει το γενικό συμφέρον. Δεν είναι δίκαιη. Δεν επιλύει το πρόβλημα της παραποίησης, αλλά ακόμη περισσότερο περιπλέκει την ισχύουσα νομοθεσία, προσπαθώντας να διευθετήσει το περιεχόμενο του διαδικτύου. Προσπαθεί να περάσει από το παράθυρο κάτι που είχε σπρώξει έξω από την πόρτα αυτό το Ευρωκοινοβούλιο με την έγκριση τον Απρίλιο του 2007 σε πρώτη ανάγνωση τη οδηγία. για την παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων και την ε, εξισορρόπηση της επιβαλλόμενης ποινής. Δεν μπορούμε λοιπόν να προστατεύσουμε το πνευματικά, τα πνευματικά δικαιώματα στο διαδίκτυο χωρίς να λάβουμε υπόψη και το δικαίωμα προστασίας του ιδιωτικού βίου και άλλα ατομικά δικαιώματα. Ολοκληρώνω λοιπόν. Ας σκεφτούμε τι πορεία μπορούμε αυστηρώς να ακολουθήσουμε και με πειθαρχία προκειμένου να δούμε το περιεχόμενο του διαδικτύου με έναν τρόπο που να μας επιτρέψει να πετύχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε. Πνευματική κάλυψη αλλά και προστασία της πολιτιστικής ποικιλότητας. Η συμφωνία ΑΚΤΑ δεν προσφέρει λύσεις ε, ως προς το θέμα αυτό και όσοι έχουν παρακολουθήσει την εξέλιξη του θέματος τα τελευταία χρόνια ξέρει ότι τελικά η τοποθέτηση του Κοινοβουλίου μας σε σχέση με αυτό που τώρα είναι στα χέρια μα και προτείνεται είναι πολύ διαφορετική. Ευχαριστώ. Έξι συνάδελφοι έχουν ζητήσει το λόγο. Ο κύριος Γκρόμπτσικ. Ευχαριστώ. χαιρετίζω τους ε, συναδέλφους. Χαίρομαι που μπορούμε να κάνουμε αυτή την ε, ανταλλαγή στην ε, Επιτροπή Ήτρε και χαίρομαι πολύ που μπορώ να πω κάτι σχετικά με την Συμφωνία Άκτα η οποία έχει δημιουργήσει πολλές αντιπαραθέσεις σε πολλά σημεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πολλά ελέγχθησαν πολύ σωστά. Όπως άλλωστε και πολλά πολύ σωστά είπε η ε, η συγκήτρια. Θέλω να αναφερθώ εδώ στις κοινωνικές πτυχές ε, του προβλήματος, διότι αν κοιτάξουμε ε, το πρόβλημα λαμβανόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει μία προστασία των πληροφοριών και της πρόσβασης και αυτό αναφέρεται στην ελευθερία ε, της διατυπώσεως ε, γνώμης και του λόγου. Ε, γι' αυτά χρειαζόμαστε πλήρη ασφάλεια για να μπορέσει να εξασφαλιστεί και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Η Πρέπει λοιπόν να φροντίσουμε να μην υπάρξει μία καταστροφή και αυτό είναι κάτι το οποίο έχουν αναφέρει πολλές πολιτικές ομάδες. Αυτό που δεν βλέπουν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο το βλέπουν οι άνθρωποι οι οποίοι ερωτούνται και βλέπουμε στις δημοσκοπήσεις ότι έχει υπάρξει μια μεγάλη κίνηση η οποία δημιουργήθηκε ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1990 από την Ανατολική Ευρώπη και το θέμα αυτό είναι πολύ σημαντικό και πολύ αμφιλεγόμενο. Η κίνηση η οποία δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1990 ουσιαστικά είναι η ίδια η οποία, την οποία να αντιμετωπίζουμε τώρα. Δηλαδή έχουμε πάρα πολλούς ε, πολίτες οι οποίοι διαδηλώνουν κατά αυτής της συμφωνίας που θεωρούν ότι περιορίζει την ελευθερία εκφράσεως του λόγου. Και εδώ βλέπουμε ότι με διάφορες μορφές υπάρχουν περιορισμοί στην ελευθερία του λόγου. και γι' αυτό και το σύστημα που είχε οικοδομηθεί μέχρι του δεν απέτυχε. Πρέπει να ξέρουμε σε τι κόσμο πρέπει να μιλούμε ε, εάν ε, κοιτάζει κανείς ε, το, τη δομή της κοινωνίας και τις απόψεις που έχουν εκφράσει οι πολίτες βλέπουμε ότι έχουν εκφραστεί διάφορες γνώμες οι οποίες περιορίζουν την ελευθερία του λόγου. Ευχαριστούμε. Η κυρία Τροτμάν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μα τα παρουσίασε πολύ καλά η συγκεκριά μα και οι σκιώδει συγκεκριτέ που πήραν ω τώρα το λόγο τα θέματα αυτά. Απλώ εγώ θέλω να θίξω και να σταθώ σε κάποια σημεία για το κείμενο τη συμφωνία. Πρώτον, συγκεκριμένο ζήτημα σε σχέση με την ε, τοποθέτηση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου εάν υπάρχει ασύμβατο μεταξύ του κειμένου τη Συμφωνία Άκτα και του κοινοτικού κεκτημένου. Θα πρέπει να αλλάξει ενδεχομένω το ευρωπαϊκό δίκαιο για να συμμορφωθούμε με το κείμενο αυτή τη διεθνού συμφωνία. Είναι καθοριστικό ζήτημα και πρέπει να απαντηθεί. Από την αρχή των όλων διαπραγματεύσεων είναι κάτι που το έχουμε στο νου μας. Το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει απόφαση λέγοντας σε ποια σημεία εντοπίζεται το ασύμβατο και πώς θα περιοριζόταν ή θα παρακολιόταν η προστασία του κοινοτικού δικαίου πάντως για την ευθύνη των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο. Υπάρχει διαρκής αναφορά στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με διαφορετικές οδηγίες. Το θέμα της ευθύνης είναι κάτι το οποίο έχει καθοριστεί. Δεν είναι υπεύθυνοι που ε, κάνουν πλέγηση στο διαδίκτυο. Ε, στα ισχυρά κείμενα αυτό που βλέπουμε είναι ότι η αρχή της μη ευθύνη όμως πλέον αμφισβητείται σε ό,τι αφορά τις ποινικέ κυρώσεις. Η Συμφωνία Άκτα εισάγει την ε, αρχή των, ε, της επιβολής κυρώσεων κατά των όσων παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα. Αυτό μπορεί να αφορά και ιδιώτες λοιπόν που χρησιμοποιούν παραποιημένο περιεχόμενο. Ακόμη και εν αγνία τους. Επιπλέον, η Συμφωνία Άκτα επιτρέπει να εξετάζονται οι προσωπικές αποσκευές των ε, ταξιδιωτών. Δηλαδή και τα MP3 και οι υπολογιστές. Ε, πώς θα βεβαιωνόμαστε ότι ένας επιβάτης δεν θα διωχθεί ποινικά για ένα τραγούδι που παρανόμως κατέβασε από το ίντερνετ λόγω χάρη. Για το περιεχόμενο του διαδικτύου λοιπόν και με την κάλυψη της καταπολέμησης της παραβίασης των πνευματικών δικαιωμάτων ε, βλέπουμε να καλύπτεται και το θέμα των παραποιημένων φαρμάκων, ένα γενώσιμο φάρμακο. Ένα πραγματικό φάρμακο που έχει εμπορευματοποιηθεί γιατί έχει λήξει η σχέση του διπλώματο ευρεσιτεχνία, οπότε δεν καλύπτεται από πνευματικά δικαιώματα, είτε γιατί ένα κράτο έχει ανάγκη να παράγει γενώσιμα για να καλύψει υγειονομικέ ε, ανάγκες. ανάγκε. Η δεύτερη αυτή περίπτωση ήδη καλύπτεται από τι συμφωνίε TRIP. Όμω η συμφωνία ACTA περιορίζει την ευελιξία των συμφωνίων TRIP και μεταχειρίζεται τα γενώσιμα φάρμακα σαν να ήταν παραποιημένα. Αυτό είναι πρόβλημα. Είναι πρόβλημα διότι υπάρχει αλλαγή ω προς τη νομική θεώρηση του ζητήματος. Πιστεύω λοιπόν ότι τα διαφορετικά αυτά σημεία εγείρουν ευρύτερο ζήτημα για την ισορροπία του όλου κειμένου. Από τη μια θέλουμε την νόμιμη προστασία των κατόχων των δικαιωμάτων, αλλά από την άλλη, όπως αυτά το είπε και ο συνάδελφός μας, την προστασία των ε, δημόσιων ελευθεριών. Διαπιστώνω ότι η συζήτησή μας και οι αντιδράσεις μας ε, στο κοινό, αλλά και οι συζητήσει στην ε, Επιτροπή μας, θέλουν να επιστρέψουμε σε μια βαθμιαία σταδιακή προσέγγιση, αλλά δεν έχουμε βρει θεμελιώδεις απαντήσεις που απαιτούνται για το κείμενο αυτό. Αυτό με συγχωρείτε πρόεδρε, για να ολοκληρώσω θεωρώ ότι είναι σφάλμα. Είναι πολύ δύσκολο βεβαίω να προσεγγίζει κανείς προβλήματα που ταυτόχρονα έχουν τόσε πολλέ προεκτάσει για του πολίτε, τι δημόσιε ελευθερίε του, την ελευθερία έκφρασή του, τη δυνατότητα πρόσβαση στα φάρμακα, τη δυνατότητα πρόσβαση στο πολιτιστικό περιεχόμενο, την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων. Είναι πολύ δύσκολο όλα αυτά να τα αντιμετωπίσουμε μόνο με ποινικέ κυρώσει και με κείμενα τα οποία από νομική άποψη παραμένουν προβληματικά, διότι δεν ορίζονται θετικά στο δίκαιο. Όταν συζητούμε με ε, εμπειρογνώμονε τη πνευματική ιδιοκτησία, ακριβώ αυτή είναι η αδυναμία τη Διεθνού Συμφωνία Άκτα. Και πρέπει τέλο να διαπιστώσουμε ότι η Επιτροπή Αναφορών μόλι έλαβε μία καταγγελία με περισσότερες από 2.400.000 υπογραφές, οπότε καλό θα ήταν να σκεφτούμε πόσο μεγάλη είναι η συσπήρωση των πολιτών, οι οποίοι παρακολουθούν το έργο μας και θα κοιτάξουν τι ακριβώς θα αποφασίσει το Κοινοβουλίο μας με μεγάλη προσοχή. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την κυρία Τροτμάν. Ο κύριος Μπαλτσίτης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι η συμφωνία αυτή είναι από τα λίγα έγγραφα που γνωρίζει τόσο αντιφατική υποδοχή στην κοινωνία. Το 2010 εμείς οι σοσιαλιστές είχαμε τελείως διαφορετική άποψη για αυτό το κείμενο. Δεν μας ακολούθησαν και τώρα πάλι για τα ίδια θέματα συζητάμε δύο χρόνια αργότερα στην Επιτροπή μας. Η συγκήτρια έχει πολύ μεγάλες επιφυλάξεις και ανησυχίες, τις εξέφρασε ήδη. Για τους ορισμούς ε, που είναι πολύ ευρύς και μπορεί να οδηγήσουν σε παρεξηγήσεις και παρερμηνίες η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων είναι σεβαστή, αλλά δεν θα πρέπει να υπονομεύει το στόχο μας και τα θέματα που μας απασχολούν σήμερα, που είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας στην Ευρώπη. Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει πολλές χώρες του κόσμου, αλλά ξέρει την Κίνα και την Ινδία, που δεν συμμετέχουν, γιατί δεν θέλησαν οι ίδιες να συμμετάσχουν. Και τώρα εμείς καλούμαστε να πούμε ένα ναι ή ένα όχι. Εγώ θα έλεγα ότι ε, δεν είναι όριμη ε, για έγκριση ακόμα η συμφωνία και θα πρέπει να το διατρανώσουμε αυτό ως Επιτροπή. Λέμε λοιπόν όχι. Ευχαριστούμε κυρία Παντιέγου. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες και τις εισηγήτριες και των υπολείπων ομιλητών, γιατί πιστεύω ότι εδώ με την ΑΚΤΑ έχουμε το εξή πρόβλημα. Και είναι πρόβλημα από γεννησιμιού της. Ε, ανακατεύουμε τα πολιτιστικά αγαθά της επικοινωνίας, της πληροφόρησης με τα καταναλωτικά αγαθά. Δεν μπορούμε να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε τη μάχη κατά της πειρατείας και κατά των απομιμήσεων και των αντιγραφών, αλλά δεν είναι η ίδια μάχη για τα πολιτιστικά αγαθά και με τα συνήθη καταναλωτικά αγαθά. Τι να κάνουμε όμως έτσι μας προέκυψε η συμφωνία. Έτσι όπως έχει γίνει όμως, το μόνο που μας απομένει ως λύση είναι το εξής. Από την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου το λέγουν και εκείνοι. Να απευθυνθούμε στο δικαστήριο για να αποφανθεί εάν παραβιάζει η συμφωνία τα θεμελιώδη δικαιώματα και αν συνάδει με την κοινοτική ε, νομολογία και δικαιοδοσία. Το μόνο που μπορούμε εμείς ε, να πούμε στη συμφωνία είναι ναι ή ένα όχι, χωρίς τροπολογίες. Οπότε γίνεται μια πρόταση να κάνουμε μια μεταβατική, μια προσωρινή έκθεση, να μιλήσει το Κοινοβούλιο, να πει τι θέλει να περιλαμβάνει αυτή η συνθήκη και τι να μην περιέχει. Είναι η μόνη διέξοδος που έχουμε για να προχωρήσουμε θα προσπαθήσω και εγώ από τη δική μας Επιτροπή να συμμετέχω στην εκπόνηση αυτής της έκθεσης στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου ακριβώς για να εκφράσουμε και τα δικά μας μελήματα. Και ένα τελευταίο, υποθέτω ότι το γνωρίζετε, ακριβώς αυτή την Πέμπτη μεθαύριο στις 3 έχουν εργαστήρι στην Ίντα για το ΑΚΤΑ. Τρεις η ώρα την Πέμπτη το απόγευμα ε, μπορούμε να πάμε εκεί να συμμετέχουμε και να ακούσουμε και πολλά ενδιαφερόμενα μέρη. Ευχαριστώ. Grazie. Ευχαριστούμε κυρία Τσικάου. Uh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα συμφωνήσω με τους συναδέλφους που θεωρούν ότι η συμφωνία ΑΚΤΑ στην τωρινή της μορφή δεν μπορεί να εγκριθεί ακόμη. Θέλω να επιρρώσω τα επιχειρήματα που ήδη ακούσαμε, διότι το άρθρο 27 της συμφωνίας, το σημείο 1, στο πρώτο εδάφιο, προβλέπει μέτρα που θέλουν να αποτρέψουν κάθε είδους παραβίαση, δηλαδή μέτρα αποτρεπτικά για κάθε είδους μελλοντική παραβίαση. Δεν ορίζεται όμως αυτή η αποτροπή θα μπορούσε να είναι και καταχρηστική χρήση. Ε, στο τέταρτο εδάφιο του 27, του άρθρου 27 και πάλι, λέγεται ότι οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να παράσχουν στον κάτοχο δικαιωμάτων πληροφορίες προκειμένου να εντοπίζεται ο κάτοχος ενός λογαριασμού. Το κείμενο αυτό δημιουργεί παρανοήσεις ό,τι αφορά και την, το σεβασμό των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών. Να θυμίσω σε όλους τους συναδέλφους της Επιτροπής Ήτρε ότι όταν συζητήσαμε τη δέσμη μέτρων για τις τηλεπικοινωνίες και μάλιστα το συζητούσαμε δυόμιση χρόνια αυτό αν θυμάστε καταλήξαμε σε διαιτησία διότι το κομβικό σημείο του όλου ζητήματος η βασική συζήτηση είχε να κάνει ακριβώς με τα δικαιώματα των πολιτών το Κοινοβούλιο επέμεινε, έδωσε μάχη ώστε να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών. Το Κοινοβούλιο επέμεινε να μην υπάρξει ούτε διακοπή παροχής υπηρεσιών από κάποιον παρέχοντα λόγω απουσία δικαστική απόφαση και προκειμένου να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα των πολιτών. Για άλλη μια φορά, αυτή η πρόληψη δεν ορίζεται παρκώ. Μπορεί δηλαδή μια αρχή να ζητήσει από έναν παροχέα πληροφοριών να δώσει πληροφορίε προκειμένου να εντοπίσει έναν συνδρομητή, έναν κάτοχο λαγαριασμού. Όλα αυτά αντιφάσκουν με την ισχύουσα ευρωπαϊκή νομοθεσία και πλήττουν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών. Ήθελε να επιστήσω την προσοχή σας στο άρθρο 14.2 επίσης. Στο δεύτερο εδάφιό του, το άρθρο αυτό ορίζει ότι ένα μέρος μπορεί να αποκλείσει μικρές ποσότητες μη εμπορευματοποιημένων προϊόντων που βρίσκονται στις αποσκευές ταξιδιωτών. Τι θα πει αυτό, μπορεί να αποκλειστούν θα μπορούσε να αποκλείσει και να μην αποκλείσει δηλαδή. Τα πάντα εξαρτώνται από την απόφαση του εν λόγου μέρους, του εν λόγου ατόμου. Μπορεί να καταλήξουμε σε καταχρήσεις. Οι αποσκευές των ταξιδιωτών, των επιβατών μπορεί να ελέγχονται στο αεροδρόμιο λόγου χάρη, στους σταθμούς, στους υδροδρομικούς σταθμούς, για να δει κάποιος αν το θέλει, κατά πόσον περιέχουν ή όχι μη εμπορικά αγαθά. προϊόντα που μπορεί να είναι να αποτελούν μάλλον, να συνιστούν παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Να θυμίσω ότι στις 24 Νοεμβρίου του 2010 το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε μια σειρά από ψηφίσματα. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών του Ευρωκοινοβουλίου, η ομάδα των Φιλελευθέρων, η ομάδα Γκουε, η ομάδα των Πρασίνων ενέκριναν, μάλλον εξέφρασαν την ανησυχία τους σε σχέση με το πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις για τη Συμφωνία Άκτα. Θεώρησαν ότι απειλούνται τα δικαιώματα των πολιτών ε, βάσει τη συμφωνία αυτή και δυστυχώ αυτά τα ψηφίσματα δεν εγκρίθηκαν. Εγκρίθηκε ένα ψήφισμα που ε, στηριζόταν από το ΕΛΚ το οποίο ε, είναι υπέρ τη συμφωνία ΑΚΤΑ και αυτό αναφέρεται και στο προήμιο. Να καταλήξω σε δύο σημαντικά συμπεράσματα. Η συμφωνία ΑΚΤΑ θα υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη. Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν ήδη προσυπογράψει στη συμφωνία. Θα ήθελα λοιπόν να θέσω το εξή ερώτημα προ του νομικού εμπειρογνώμονε. Α φανταστούμε ότι η συμφωνία αυτή απορρίπτεται από το Ευρωκοινοβούλιο. Τι θα γίνει με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών σε χώρε μέλη που έχουν ήδη υπογράψει τη συμφωνία και την έχουν εγκρίνει. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι δεν υπάρχει απλώς μια αναφορά. Θα μπορεί να υπάρξει μια ολόκληρη πρωτοβουλία των ε, Ευρωπαίων πολιτών που να έχει να κάνει με την Συμφωνία Άκτα στο μέλλον. Νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καταψηφίσουμε τη Συμφωνία Άκτα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν σεβόμαστε τα, δικαιώματα, τα πνευματικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε ήδη κεκτημένο που αφορά την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων, όμω επιθυμούμε μια συμφωνία η οποία να βελτιωμένη και να ε, μεταχειρίζεται με τρόπο ισοδύναμο του Ευρωπαίου πολίτε. Ευχαριστούμε, ο κύριο Κέλλη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Υπάρχει μια σαφή στάση να συμφωνούν μεταξύ του όλοι ε, οι ομιλητέ σήμερα. Κανεί δεν είναι ευχαριστημένο με όσα προτείνονται. Και φαντάζομαι ότι η συγκήτρια σωστά είπε ότι είναι κάπως βιαστικά όλα αυτά. Προσπαθούμε να καταφέρουμε περισσότερα από όσα μπορούμε. Και αυτό πολύ αγχώνει και δυσκολεύει το κοινό. Όλοι θα ήταν υπέρ μιας τέτοιας συμφωνίας, διότι όλοι θέλουμε να περιοριστεί η παραποίηση προϊόντων. Σίγουρα πλήττεται το ετήσιο ΑΕΠ και βεβαίως τα τελευταία 7 χρόνια ήταν πολύ σημαντικές οι επιπτώσεις από την ε, παραποίηση. όμως πρέπει να περιοριστούμε στη συμφωνία άκτα και να δούμε ζητήματα όπου μπορεί να εμπλέκονται ε, παρανομούντες Αυτοί που διαπράττουν πειρατεία. Μην ξεχνάμε κάποιες φορές εμπορεύματα από την Κίνα που είναι παραποιημένα. Να το αντιληφθούμε αυτό, διότι σε αυτή τη φάση είναι πολύ αυτοί που ανησυχούν για την ελεύθερη κυκλοφορία στο ε, διαδίκτυο, για τους κανόνες προστασίας προσωπικών δεδομένων. Εδώ η συζήτηση έχει μετατοπιστεί από, την, ε, από το τι γίνεται με τη Συμφωνία Άκτα. Και σκεφτόμαστε την παραποίηση προϊόντων. Αυτό θα έπρεπε να είναι ο βασικός μας στόχος. Η κυρία Μπαντία Ικουτσέτ ανέφερε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την απόφαση που αναμένεται. Όμως εδώ χρειαζόμαστε κάτι αποτελεσματικό και το χρειαζόμαστε γρήγορα. Διότι θέλουμε οι πολίτες να αντιληφθούν ότι κάτι προσπαθούμε να κάνουμε, ότι είναι δίκαιο αυτό και να τους έχουμε με το μέρος μας, όχι να τους αποξενώσουμε. Χρειαζόμαστε όμως πιο συγκεκριμένους ορισμούς και των δικαιωμάτων πραγματική ιδιοκτησία και όλων των άλλων ζητημάτων που αυτή τη στιγμή βρίσκονται επιτάπητος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Κάσπαρη. Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Το θέμα αυτό της άκτα Νομίζω ότι είναι ιδίω ένα σημαντικό θέμα όπως άλλοτε ανέφερε ο προλαλής σας διότι είναι πολύ σημαντικό αν έχουμε να κάνουμε με παραποιημένα προϊόντα και έχει δημιουργήσει ε, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην ε, κοινή γνώμη λόγω παραπληροφόρησης και κακής ενημέρωσης των πολιτών. Εκπλήσωμαι όταν βλέπω πόσο συμμετέχουν συνάδελφοι εις ε, την δημιουργία και ε, αναζωπήρηση αυτής ε, της αρνητικής κινήσεως διότι ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης και εάν δεν δεν υπάρξει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για αυτό το νομοθέτημα δεν θα ισχύσει και είναι κρίμα. Εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απορρίψει το άκτα δεν θα ισχύσει. Πρέπει λοιπόν να γνωρίζουμε ε, περί τίνος πρόκειται, δηλαδή να γνωρίζουμε ότι στην αρχή της διαδικασίας ε, πρέπει να ξέρουμε όλοι ότι ε, σαν συνομοθέτες έχουμε μεγάλη ευθύνη, πολύ μεγάλη από ό,τι θα είχαμε πριν από δύο χρόνια πριν να ισχύσει η συνθήκη της Αβώνας. Τότε μπορούσαμε να πούμε ότι δεν μας αρέσει αυτό ή εκείνο και καλούμε τους ε, υπολείπους να ακολουθήσουν τις απόψεις μας για να μπορέσει να υλοποιηθεί. Αλλά τώρα θα πρέπει να ενεργούμε με υπευθυνότητα και γι' αυτό πρέπει με ηρεμία να ελέγξουμε αυτή τη συμφωνία διότι στο ΕΛΚ δεν χρειάζεται να εξηγήσει κανείς τι σημαίνει η ελευθερία του διαδικτύου. Έχουμε πολλούς συναδέλφους στην πολιτική ομάδα οι οποίοι λόγω καταπιέσεων ε, και ε, διωγμού από την ε, κομμουνιστική, από τα κομμουνιστικά καθεστώτα της Ανατολικής Ευρώπης έχουν διωχτεί και έχουν διατυπώσει δύο γνώμη. Λοιπόν, όταν βλέπουμε επιπλέον ότι πάνω από 10.000, ότι πολλές δεκάδες χιλιάδες θέσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταργούνται λόγω μετακινήσεων κινήσεως των, ε, ε, των επιχειρήσεων όταν στα αυτοκίνητα το 70% των ανταλλακτικών τα οποία πολλούνται ε, είναι παραποιημένα και όχι, δεν προέρχονται από εκεί που αναγράφεται στην ε, συσκευασία τότε δεν μιλάμε μόνο για την ελευθερία στο διαδίκτυο αλλά για ανθρώπινες ζωές, για ανταλλακτικά αεροπλάνων διότι βλέπουμε ότι ένα 5% των ε, ανταλλακτικών αεροπλάνων είναι παραποιημένα και αυτό διακινδυνεύει κινδυνεύει ανθρώπινες ζωές. Άρα είναι θέματα για τα οποία το ΕΛΚ έχει ευαισθητοποιηθεί και έχει πει ότι δεν θα αλλάξει με την άκτα η ζωή των Ευρωπαίων στην Ευρώπη αλλά θα πρέπει ε, να υπάρχει μία γενική συμφωνία και όχι με πολλές λεπτομέρειες που πλέον ε, θα υπάρχει παραλογισμός. Ε, δεν θέλουμε επιταγές, δεν θέλουμε ή στο μέλλον οι πολίτες μας να καταπιέζονται και απλώς στις χώρες όπου επιτρέπονται τέτοιες μεθοδολογίες μπορούν να συνεχίσουν αλλά δεν θέλουμε στην Ευρώπη να ισχύσουν τέτοιες προϋποθέσεις. Η συμφωνία λοιπόν αυτή είναι ένα πρόβλημα διότι δεν συμμετέχουν η Κίνα και η Ινδία και όπως είπε και ο κύριος Κέλλη τα περισσότερα παραποιημένα προϊόντα προέρχονται από αυτές τις χώρες οι οποίες δεν συμπράττουν. Αλλά έχουμε προσπαθήσει στον ΠΟΕ και σε όλες τις διεθνείς οργανώσεις να προχωρήσουμε και να καταπολεμήσουμε τα παραποιημένα προϊόντα τα οποία διακινούνται διεθνών και τώρα υπάρχει μία ένωση και ένα συνασπισμό των χωρών που θέλουν να ισχύσει το άκτα και ακόμη και αν δούμε το πρωτόκολλο του Κιώτο και την προστασία του κλίματος αναρωτήθηκε πολύ ποτέ καλήσω ότι μπορεί να μην συμπράττουν στο πρωτόκολλο του Κιώτο οι Κινέζοι και οι Αμερικάνοι αλλά εμείς προχωρούμε ακόμη και αν οι μεγαλύτεροι ρηπαντές δεν ακολουθούν. Το ίδιο πρέπει να συμβεί και με το άκτα. Θα πρέπει να ξεκινήσουμε να ελέγχουμε με ηρεμία το θέμα αυτό και θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό που ο κύριος ε, David Μάρτιν έχει καταρτήσει μία ενδιάμεση έκθεση. Πρέπει να δούμε ε, πού μπορούμε να επιτύχουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγγυήσει ε, για τα μεταβατικά μέτρα και από τα κρατη άλλωστε. Πρέπει να δούμε πώς θα εμπλακεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και όλοι θα πρέπει να φροντίσουν να κοιτάξουν τι θέματα θεωρούμε ότι ε, είναι επικίνδυνα και πρέπει να υποβληθούν σχετικές ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τέλος όταν ε, όλες αυτές οι ερωτήσεις θα έχουν απαντηθεί θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε ε, χωρίς να κάνουμε κάτι με κλειστά τα μάτια. Ευχαριστώ που μου δώσατε χρόνο κυρία Πρόεδρε Πρόεδρε, αλλά προσπάθησα με κάθε τρόπο να διατυπώσω τις δικές μου ανησυχίες και αντιρρήσεις. Ευχαριστώ. Για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Το όνομά μου είναι Μπολορολέ και μιλώ εν ονόματι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να παρουσιάσω και να εξηγήσω αυτό το οποίο ε, είναι η άκτα Όσον αφορά την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στόχος είναι να ε, βελτιωθούν οι νομικές προδιαγραφές κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή ε, δεν θέλουμε να βελτιώσουμε το δικαίωμα προστασίας αλλά πρόσβαση στη δικαιοσύνη για να υπερασπιστούμε καλύτερα τα δικαιώματα της πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτές οι προδιαγραφές προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας ισχύουν ήδη στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα ε, το σύνολο νομοθετημάτων της και ε, η άκτα θα μπορέσει να ε, αναβαθμίσει σε διεθνές πολυμερές επίπεδο αυτά τα νομοθετήματα. Δεν θα αλλάξει κάτι στο ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο, αλλά η άκτα είναι σημαντική για τις εμπορικές συναλλαγές που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τις τελευταίες εβδομάδες η ε, κύρωση αυτής της συμφωνίας προκάλεσε πολλές συζητήσεις και πολλές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιλαμβάνεται πλήρως τις κριτικές και τις συζητήσεις όπως και τα ε, σημεία τα οποία έχουν θέσει ορισμένοι στα πλαίσια αυτά. Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνθηκε στο Ευρωπαϊκό ο δικαστήριο για να υπάρχει μία ισορροπία μεταξύ ε, των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και ε, βασικών θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί η μετάβαση αυτή να γίνει σοσκελισμένα και ήρεμα και να μην ε, διαβρωθεί από άλλα από άλλους παράγοντες. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η σημασία της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι πολύ σημαντική και δεν άπτεται μόνο της άκτα. Η άκτα είναι απλώς μία συμφωνία που αναφέρεται στην πρόσβαση προς τη δικαιοσύνη. Τίποτα παραπάνω, τίποτα παρακάτω. Η πρόσβαση αυτή στη δικαιοσύνη πρέπει να είναι εφικτή για αυτούς που έχουν δικαιώματα ή ε, τον πραγματικό κόσμο, δηλαδή για τους ε, παραγωγούς προϊόντων ε, απτών, αλλά και τους ιδιοκτήτες πνευματικής ε, ιδιοκτησίας οι οποίοι ε, συναλλάσσονται στο διαδίκτυο. Δεν έχει όμως στόχο να αμφισβητήσει τα δικαιώματα πνευματικής ε, ιδιοκτησίας ούτε την ιδέα της διακίνησης στο διαδίκτυο. Δεν είναι αυτός ο στόχος της άκτας και το τονίζω και πάλι. Euh, όπως τόνισε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι σημαντικό να γίνονται νυφάλιες συζητήσεις. Ε, η παραπομπή στο δικαστήριο τη συμφωνία αυτής για να μάθουμε αν ανταποκρίνεται και ευθυγραμμίζεται με τα θεμελιώδη δικαιώματα θα επιτρέψει στους πάντες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα διάφορα θεσμικά όργανα που ενέχονται στην νομοθετική διαδικασία να κάνουν συζήτηση. Σήμερα είναι μια πρώτη ευκαιρία. Την ερχόμενη Πέμπτη ο Επίτροπος Ντεχιόχτ θα έρθει ενώπιον της Επιτροπής ΙΝΤΑ και θα συζητήσει το ζήτημα του ΑΚΤΑ και όλα τα σημεία ε, που ε, υπευλήθησαν και σήμερα το απόγευμα. Αργότερα Τις επόμενες εβδομάδες θα συνεχιστούν οι συζητήσεις και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να μπορεί να συμμετέχει όσο γίνεται στις συζητήσεις αυτές. Τώρα για να απαντήσω πιο συγκεκριμένα σε ορισμένα θέματα που αναφέρατε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να θυμίσει ότι η Άκτα είναι ε, μια διεθνή σύμβαση, συνθήκη που προσφέρει ένα νομικό πλαίσιο. Διεθνούς δικαίου, ένα διεθνές νομικό πλαίσιο. Κατά ανάγκη λοιπόν, τα συμβαλόμενα μέρη έχουν μια σειρά επιλογών στη διάθεσή τους. Και σε αυτά τα μέρη εναπόκειται, αυτή τη στιγμή στεθεί σε ισχύ η συμφωνία να ορίσουν ποιες επιλογές επιθυμούν να εντάξουν στην ε, εσωτερική τους νομοθεσία. Σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, το πλαίσιο είναι προκαθορισμένο ήδη, υπάρχει και είναι η οδηγία E-PRED το 2004 που ακούστηκε ή και το e-commerce που ορίζει την εμπορική δραστηριότητα στο διαδίκτυο ή την οδηγία για τα πνευματικά δικαιώματα στην κοινωνία της πληροφορίας του 2001. Άρα υπάρχουν αυτά τα νομοθετήματα και το νομικό πλαίσιο στο οποίο θα λειτουργήσει η άκτα υφίσταται και δεν θα τροποποιηθεί λόγω της έλευσης αυτής της συμφωνίας. δεν προβλέπει σε καμία περίπτωση η άκτα ούτε να κόβεται το διαδίκτυο, ούτε να ε, σταματάει η σύνδεση, ούτε να υπάρχουν κάποιες ιδιωτικές αστυνομίες, όπως ακούστηκε και αυτό. Προβλέπεται μόνο η δυνατότητα να υπάρχει ένας κώδικας δεοντολογίας για να συντονίζονται οι φορείς του διαδικτύου. Υπάρχει αυτό ήδη το άρθρο 16 της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο ή 17 της εφαρμοστικής οδηγίας προβλέπεται η δυνατότητα ε, κώδικα ε, δεοντολογίας και συμπεριφοράς μεταξύ των διαφόρων ενεχομένων. Δεν σημαίνει ότι αυτό θα οδηγήσει ιδιωτική αστυνόμευση, όπως ακούστηκε είπαμε. Αλλά η άκτα θεμελιώνεται σε μια διεθνή συμφωνία που ήδη υπάρχει, η ΑΤΠΗ του 1994 και ορισμένα κράτη που αδυνατούν να ε, ενημερώσουν αυτή τη συμφωνία, να την επικυροποιήσουν στα πλαίσια του ΠΟΕ ή σε άλλα διεθνή φόρα, αποφάσισαν να βελτιώσουν τους κανόνες μέσω μιας νέας σύμβασης ε, που ονομάζεται ΑΚΤΑ. Αυτά. Ευχαριστώ. Η Πρόεδρος, ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή την παρέμβασή του. Το λόγο τώρα έχει η συγγήτρια κυρία Άντερς Ντότερ, παρακαλώ για να απαντήσει. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για ε, τη συνεισφορά τους στη συζήτηση και για τα πολλά και σημαντικά σχόλια που έκαναν. Ιδιαίτερα αυτά που αφορούσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις σχέσεις στο διαδίκτυο, αλλά και τα προβλήματα με τα εμπορικά σήματα, κοινώς μάρκες. Εγώ θα περίμενα να μας βοηθήσει περισσότερο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εμά, την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο γενικότερα. Να μας πει ε, τι μελέτες έχουν γίνει για την ισχύουσα νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το έχετε σκεφτεί αυτό, το έχετε παρακολουθήσει. Τι γίνεται με τη Συμφωνία για την οδετερότητα του Δικτύου. Τι γίνεται με την ίση μεταχείριση της κυκλοφορίας των δεδομένων και των πληροφοριών και στη διαδικτυακή αγορά υπηρεσιών. Έχουμε χρόνο όμως, μπορούμε να επανέλθουμε στη συνέχεια, να ξανακάνουμε συζητήσεις. Θα παρακαλούσα και θα εκτιμούσα πολύ αν μπορούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει και από αυτού του συγκεκριμένου. Ευχαριστώ. Πριν προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. Θα σας δώσω μία ενημέρωση σχετικά με τη συνάντηση των συντονιστών εχθές όπου υπήρξαν ορισμένες αλλαγές που έγιναν στο χρονοδιάγραμμα και θα κοινοποιηθούν στους συναδέλφους. Αποφασίσαμε για το ταξίδι στο Βραζιλία. Ε, αποφασίσαμε ότι το Μάιο θα γίνει μία δημόσια ακρόαση για τον ορίζοντα 2020 και ε, ε, θα, διαρκέσει μία ολόκληρη ημέρα και στις 8 Μαΐου θα υπάρξει μία ακρόαση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης, ε, η κυρία Τόγια καθορίστηκε σαν εισηγήτρια για την Επιτροπή και στην ε, Γκουε ανατέθηκε το πρόγραμμα ΙΤΕΡ ε, και ε, όσον αφορά την έκθεση και για τη γνωμοδότηση στο ΕΛΚ και στους πρασίνους ο προϋπολογισμός του 2013. Αυτές ήταν οι πληροφορίε που έπρεπε να σας, να σας δώσω και τώρα θα κοιτάξουμε το τελευταίο θέμα το οποίο έχουμε, Project Bond και το λόγο έχει ο κύριος Πίπερ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρόκειται για μία έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμού και απλώς γνωμοδότηση της δικιάς μας ε, Επιτροπής και με παρακάλεσε ο κύριος Λάνιεν ε, εν τη απουσία του επειδή βρίσκεται σε ταξίδι σε μία αποστολή να κάνω μία σύντομη παρουσίαση. Έχουμε ε, το πρόγραμμα αυτό και και θέλουμε να δοκιμάσουμε διάφορα μέσα κατά την περίοδο 2014-2020 έχουμε διάφορα προγράμματα ε, όσον αφορά την χρηματοδότηση και την χορήγηση κοινοτικής οικονομικής συνδρομής για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών και ενέργειας. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν κενά, διότι υπάρχουν και προγράμματα που είναι απλώς business as usual, δηλαδή τετριμένα και δεν έχουν μία άμεση σχέση με, την ε, ευρωπαϊκή, με τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής υπεραξίας, προστιθέμενης αξίας. Και ε, γι' αυτό θεωρούμε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι της γνώμης ότι δεν θα υπάρξει καμία νέα κίνηση και δεν θα ελέγξουμε κάτι προοδευτικό. Ως εκ τούτου το Κοινοβούλιο θεωρεί ότι δεν θα συμφωνήσει εις το business as usual και ε, αυτά ε, ήταν η γνώμη του κυρίου Λάγκεν. Σας ευχαριστώ για την ε, προσοχή σας. Αυτά είχα να σας πω. Ευχαριστώ τον κύριο Πίπερ. Υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να σχολιάσει αυτό το θέμα. Ο κύριος Κρόιτσμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ να είμαι σύντομος. Αυτό που πρότεινε ο κύριος Λάγκεν μας βρίσκει σύμφωνους και τον υποστηρίζουμε. Αλλά για τα ομόλογα έργων θα πρέπει να δούμε αν είναι βιώσιμα τα έργα αυτά και αποδοτικά καταρχάς. Κατά δεύτερο λόγο, να μην ενισχύσουμε έργα κύριε Πίπερ, όπως είπατε, που είναι ήδη τετριμένα και ε, συνηθισμένα, αλλά άλλα που να έχουν ευρωπαϊκή υπεραξία και είναι πολλά αυτά. Και μέσω των ομολόγων έργων μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη μόχλευση για να επιτύχουμε να προσελκύσουμε ιδιωτικά κεφάλαια. Και μετά ε, τα έργα αυτά που θα χρειαστούν τα επόμενα χρόνια να τα υλοποιήσουμε. Είναι υποδομές, είναι έργα στην ηλεκτρική ενέργεια, ε, στη διανομή φυσικού αερίου κτλ. Σε πολλούς τομείς δεν έχουμε ολοκληρώσει ακόμα την εσωτερική αγορά και μπορούμε να δημιουργήσουμε ανάπτυξη και με τα ομόλογα έργων. Γι' αυτό υποστηρίζουμε την παρούσα πρόταση και σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κέλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι ότι επιτέλους υπήρξε μία πρόοδος σε ένα θέμα το οποίο ε, επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και μερικά χρόνια και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να επιτύχουμε κάποια προστιθέμενη αξία και να μπορέσουμε ε, να ε, λύσουμε το θέμα της οικονομικής κατάστασης διότι πρέπει όχι μόνο να διερευνήσουμε το θέμα αλλά και να το δοκιμάσουμε κατά τρόπον ώστε να υπάρξει δυνατότητα να υπάρχουν ορισμένα προγράμματα τα οποία θα ισχύσουν και να προσπαθήσουμε το 2020 ε, να έχει στόχους οι οποίοι μπορούν να υλοποιηθούν διότι αυτό είναι το βασικό και αν το επιτύχουμε τότε θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε ένα νέο σύστημα το οποίο θα μπορεί και να χρηματοδοτηθεί και να ισχύσει. Ενώ, εάν μιλάμε για business as usual και δεν υπάρχει προστιθέμενη αξία, θα έχουμε αποτύχει. Οπότε, το πρόγραμμα και η στρατηγική για το 2020 ή όπως και να ονομάζεται είναι κάτι το οποίο πρέπει να προωθήσουμε με κάθε τρόπο με τον οποίο μπορούμε. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη και εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις το λόγο έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όχι. Η κυρία Χέρτσοκ όμως them, please. Uh, sorry, Chairman, being late, but we discussed the same subject in the budget. Ε, ναι, συζητούμε το ίδιο θέμα στην Επιτροπή ε, Προϋπολογισμών, συγγνώμη. Ε, είναι ενδιαφέρον να δει κανείς και στις άλλες επιτροπές πώς το συζητούν και ε, ε, κάθε επιτροπή το βλέπει από το δικό της πρίσμα βεβαίως. Οι δύο επιτροπές που γνωμοδοτούν έχουν συντάκτες γνωμοδότησης από το ΕΛΚ και οι δύο, αλλά η προσέγγιση τους είναι πολύ διαφορετική. Ο κύριος Κάντσαν ζητάει ακόμα πιο ριζική λύση για τα, ομόλογα, τα ευρωομόλογα. Από τη γνωμοδότησή σας έχω την αίσθηση ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τα πιλωτικά προγράμματα. Θα πρέπει να καταλάβουμε όμως ότι έχουμε μόνο 18 μήνες ε, πριν τις νέες δημοσιονομικές προοπτικές και κατά τη διάρκεια αυτών των 18 μηνών θα πρέπει να κάνουμε ε, όλα αυτά από τα πιλωτικά προγράμματα με τις συνέπειές τους για να βγάλουμε και τα συμπεράσματά μας. Θα πρέπει σε τόσο λίγο χρόνο να επικεντρωθούμε σε ένα τελείως νέο ε, σύστημα αν θέλουμε να επιτύχουμε. Και σίγουρα θα κάνουμε και κάποιες τροπολογίες στην έκθεση του κυρίου Λάγκεν. Δεν καταλαβαίνουμε γιατί στην τροπολογία 2 θέλει να περιορίσει τα ομόλογα ε, έργων για τα έργα υποδομής και μόνο. Ενώ υπάρχουν και άλλα έργα που μπορεί να είναι στην ανανεώσιμη ενέργεια ή στα αποκεντρωμένα συστήματα ενέργειας. Ε, δεν καταλαβαίνουμε γιατί θα πρέπει να το περιορίσει οπωσδήποτε στα έργα υποδομής. για ε, το μακροπρόθεσμο, όχι τα πιλωτικά προγράμματα τώρα, θα πρέπει να παραμείνει αυτό ανοιχτό. Είναι από τα σημαντικά μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Έτσι δεν είναι. Έχουμε προβλήματα με αυτή την τροπολογία. Γενικά συμφωνούμε όμως με τον εισηγητή ότι αυτό το μέσο είναι μια προσθήκη. Δεν έρχεται να αντικαταστήσει ούτε τη συνεισφορά των κρατών μελών, ούτε του κοινοτικού προϋπολογισμού, ε, ούτε τίποτα άλλο. Είναι προσθήκη σε εκείνα τα έργα που δεν είναι ε, συμφέροντα από πλευράς εμπορικής. Και στην Επιτροπή Προϋπολογισμών τα γνωρίζουμε πολύ καλύτερα αυτά τα θέματα. Και α είμαστε ειλικρινεί, α μην γελιόμαστε. Τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια που τουλάχιστον συμμετέχω εγώ στο Κοινοβούλιο, οτιδήποτε προσπαθήσαμε ε, να κάνουμε για να εξυγχρονιστεί η υποδομή σε όλη την Ευρώπη, απέτυχε θυμάστε το στρατηγικό τεχνολογικό πρόγραμμα για να σας αναφέρω ένα και μόνο. Και θα πρέπει να καταλάβουμε ότι αν δεν ανανεώσουμε ε, τις υποδομές και στην ενέργεια και στις τηλεπικοινωνίες, η επόμενη γενιά σε 10 χρόνια θα αντιμετωπίσει πρόβλημα. Είναι πολλά αυτά που διακυβεύονται εδώ για να αποτύχουμε. Δεν επιτρέπεται και γι' αυτό νομίζω αυτό θα πρέπει να είναι ο, ο γνώμονας ε, στην εργασία μας. Είμαι σίγουρη ότι θα βρούμε μια λύση για να υποστηρίξουμε πιλωτικά προγράμματα και να προχωρήσει αυτό όχι μόνο για τις υποδομές ενέργειας, όχι μόνο για τα έργα υποδομής δηλαδή, αλλά και στην ενέργεια και ε, στις τηλεπικοινωνίες. Θα κάνουμε και τροπολογίες αντίστοιχα και ελπίζω να συμφωνεί και ο εισηγητής μαζί μας σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστώ. Ωραία, δεν υπάρχουν άλλες παραβάσεις. Μήπως ο κύριος Πίπερ θέλει κάτι να πει ακόμη. Ευχαριστώ. Ε, είμαι επιφυλακτικός σχετικά με την πρόταση ε, της συναδέλφου Χέρτσοκ για να περιλάβουμε την πρότασή της διότι όντως θα πρέπει να υπάρχει ένας πιλωτικός χαρακτήρας και να υπάρξει μία προστιθέμενη αξία. Είναι μία προσθήκη την οποία θα πρέπει να εξετάσουμε και να συμφωνήσουμε. Ευχαριστώ κύριε Πίπερ. Με αυτό έχουμε τελειώσει τη συζήτηση αυτή. Ο χρόνος για την υποβολή των ε, τροπολογιών είναι μέχρι τις 5 Μαρτίου το μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν ε, καλύψει όλη την ημερήσια διάταξη και η επόμενη συνεδρίαση θα είναι 29 και 20 Μαρτίου στις Βρυξέλλες. Ευχαριστώ και καλό βράδυ.